Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Χαιρετώ λοιπόν, είσαστε υπεύθυνο για την βιομηχανική πολιτική. Έχουμε σε πολλές περιπτώσεις συζητήσει το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής, λέγοντας ότι πρέπει να ξαναδούμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό μας, να ξαναδούμε ποια είναι τα αδύναμα και τα δυνατά σημεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φερχόγγεν που ήδη από την αρχή της θητείας αυτής της Επιτροπής είστε διαθέσιμος και θελήσατε να έρθετε και να μας μιλήσετε για διάφορα θέματα που αφορούν την πολιτική της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η Επιτροπή αυτή. Θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ διότι αναλάβατε την Προεδρία και βεβαίως πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα, ένα θέμα που αφορά την βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι η βιομηχανική πολιτική είναι ένας νέος τομέας γιατί παλαιότερα η βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, αν θέλετε, μια προστατευτική και παρεμβατική ε, προσέγγιση. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει πλέον. Η δική μας προσέγγιση έχει αλλάξει. Θέλουμε μια δυνατή, σύγχρονη βιομηχανική πολιτική, η οποία να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στους τομείς που χρειάζεται στον τομέα των υπηρεσιών και σε όλους τους άλλους τομείς. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις, ένα πλαίσιο το οποίο να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία από το προηγούμενο καλοκαίρι, από πέρσι το καλοκαίρι, έχει μπει σε μία από τις πιο σοβαρές οικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών και 10 και η παραγωγή βιομηχανικής στην Ευρώπη βρίσκεται σε συνεχή πτώση. Το τελευταίο τετράμινο, ε, τρίμηνο, συγγνώμη, αυτή η πτώση σταθεροποιείται. Παρόλα αυτά, είμαστε σε επίπεδα του 97 πλέον. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι από εδώ και πέρα χρειάζονται ανακατατάξεις, προσαρμογές, θα υπάρξουν νεύσεις και εξαγορές εταιριών, αλλά δυστυχώς θα υπάρξουν και επιχειρήσεις που θα εξαφανιστούν από την αγορά. Και αυτό δυστυχώς πλήττει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια θετικά ε, σημεία σε αυτή την κρίση. Η εσωτερική αγορά έδειξε εξαιρετική σταθερότητα. Δεν επλήγει όπως θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Και νομίζω ότι από κοινού πετύχαμε εμείς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να αποφύγουμε μία ελεύθερη πτώση, να αποφύγουμε προστατευτισμό και εθνικισμό, που είναι οι φυσικές τάσεις όταν υπάρχει οικονομική κρίση. Πετύχαμε επίσης και προγράμματα, να αναπτύξουμε προγράμματα ανάκαμψης, κάτι που πραγματικά ξεκίνησαν, το είδαμε αυτό σε πολλές χώρες, όχι τα παραδοσιακά προγράμματα ενίσχυσης μέσω επιδόσεων, αλλά προγράμματα ανάκαμψης τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους και πιο μακροπρόθεσμους στόχους με επενδύσεις που πραγματικά στο μέλλον θα βοηθήσουν μέσω της έρευνας, ανάπτυξης και εξυγχρονισμού των υποδομών να βοηθήσουν την οικονομία μας να στραφεί προς το μέλλον. Υπάρχουν σήμερα ιδιαίτερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες αγοράς της Ευρώπης, δυνατότητες ανάπτυξης. Υπάρχουν ακόμα αγορές τις οποίες η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται και να είναι έντονη. Χρειάζεται λοιπόν να δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στα νέα προϊόντα, κάτι που μπορεί να μας ανοίξει και νέες αγορές. Τώρα, τα αρνητικά σημεία. στον τραπεζικό τομέα η κατάσταση κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι πίσω μας. Θα δούμε βεβαίως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το θέμα αυτό. Η χρηματοδότηση ακόμα δεν είναι στα επίπεδα που θα θέλαμε ή που θα έπρεπε. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν οι προσπάθειες για καλύτερη ροή των κονδυλίων. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα τελευταία χρόνια αποκομίσαμε κάποια διδάγματα. Υπήρξαν τομείς όπου αναγνωρίζουμε ελλείψεις. Πολύ συγκεκριμένα θα ήθελα να πω ότι για να είναι ανταγωνιστική η βιομηχανία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είμαστε πολύ ισχυροί στον τομέα της καινοτομίας. Και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ επίγον. Θα πρέπει να στηρίξουμε όχι μόνο την οικονομία που βασίζεται στη γνώση, αλλά και την οικονομία που βασίζεται σε πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, low carbon industry, και τομείς που επιβάλλουν περαιτέρω επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Η Επιτροπή λοιπόν Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς αυτούς. Η πολιτική στον τομέα της καινοτομίας. Βεβαίως και έχουν γίνει σημαντικά βήματα το τελευταίο καιρό, αλλά το συνολικό αν θέλετε ε, περιβάλλον δεν είναι ικανοποιητικό, δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε. Και πρέπει πραγματικά να βρούμε ποια είναι τα αδύναμα σημεία και να τα ενισχύσουμε. Υπάρχει πολλής κατακαιρματισμός, υπάρχει γραφειοκρατία, δεν υπάρχει κεντρική αντιμετώπιση των σχεδίων. Και βεβαίως συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα στην διάθεση, στην αγορά, στην εμπορική διάθεση των προγραμμάτων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Νέα πρότυπα, νέα πολιτικά εργαλεία που για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν σε ένα πακέτο στρατηγικών μέτρων και ακριβώς αυτό θα κάνουμε τα επόμενα έξι χρόνια με ε, μια ευρωπαϊκή πράξη για την καινοτομία, μια νέα φάση, ένα πακέτο μέτρων κάτι που θα ξεκινήσουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά επίγον να συμπεριλάβουμε αυτά τα μέτρα στις μελλοντικές μας πολιτικές αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστές Ξέρετε τι κάνουν οι Αμερικανοί. Ο πρόεδρος Ομπάμα ανακοίνωσε την Αμερικανική νέα στρατηγική στον τομέα της καινοτομίας τον Αύγουστο. Η αμερικανική και οι δική μας στρατηγική έχουν κάποια κοινά σημεία. Οι τεχνολογίες κλειδιά, όπως τις ονομάζουμε, key technologies, είναι οι τεχνολογίες του 21ου αιώνα. Αυτές που θα έπρεπε τουλάχιστον να επικρατήσουν και να αναπτυχθούν στον 21ο αιώνα. Και όταν λέω να επικρατήσουν δεν εννοώ ότι μόνο εκεί θα επενδυθούν ε, κονδύλια σε αυτού του είδους την έρευνα, αλλά θα πρέπει στην παραγωγή να χρησιμοποιούνται αυτές οι νέες τεχνολογίες. Πριν από λίγες εβδομάδες προετοιμάσαμε κάποιες προτάσεις για αυτές τις ε, τεχνολογίες κλειδιά οι οποίες καταρχήν θα πρέπει να εντοπιστούν, ε, τεχνολογίες που έχουν στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή πολιτική, όπως οι νανοτεχνολογίες, νάνο και μικροηλεκτρονική, νέα υλικά, φωτονική και βεβαίως όλος ο τομέας της βιοτεχνολογίας. Πρόκειται για 4-5 τομείς, οι οποίοι θεωρούνται τομείς τους οποίους έχουμε εντοπίσει και τους οποίους θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω. Η πολιτική μας, όπως είπα και στην αρχή, δεν έγκυται σε μία άμεση επέμβαση, παρέμβαση σε τομείς ή σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Σκοπός μας είναι να θέσουμε το πλαίσιο και η γενική κατεύθυνση είναι καινοτομία με εκπαίδευση, με έρευνα και ανάπτυξη, με νέες υποδομές, σύγχρονες υποδομές, οι ευρυζωνικές τεχνολογίες παραδείγματος χάριν και το θέμα της εξωτερικής διάστασης της ανταγωνιστικότητάς μας, πώς δηλαδή στο μέλλον οι εμπορικές μας συναλλαγές θα πρέπει να διευθετηθούν με μια ολόκληρη σειρά νέων ε, συμβάσεων οι οποίες όπως ξέρετε είναι εν εξελίξη εκκρεμούν ή θα υπογραφούν από την επόμενη εβδομάδα κιόλας νέες συμφωνίες για το παγκόσμιο εμπόριο και τις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν την Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσω αυτών των νέων συμφωνιών που όχι μόνο θα διευκολύνουν την κατάσταση για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας, αλλά την ίδια ώρα θα αφήσουμε καλύτερη πρόσβαση στα προϊόντα άλλων χωρών και υπήρων και τα δικά μας προϊόντα θα μπορούν να διεισδύσουν καλύτερα σε νέες αγορές. Θα πρέπει επίσης τα επόμενα χρόνια να ασχοληθείτε ιδιαίτερα με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πνευματικών δικαιωμάτων και το θέμα αυτό πρέπει να πω ότι δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε. Δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη αρκετή πρόοδος ούτε στο copyright, ούτε στο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρωσιτεχνίας, κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί ένα εμπόδιο και ένα μειονέκτημα για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και θα στραφώ τώρα σε μια έκθεση πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Σήμερα υπάρχει η σαφής ανάγκη όλα τα πολιτικά εργαλεία που διαθέτουμε να διευκολύνουν την πρόσβαση στα λεγόμενα στρατηγικά προϊόντα, στρατηγικές πρώτες ύλες. Αυτές που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, που δεν είναι διαθέσιμες στην Ευρώπη και οι οποίες είναι απαραίτητες εκεί που η στην αγορά, η διείσδυση στην αγορά είναι ακόμα δύσκολη και δεν είναι εύκολο να διαπραγματευτεί κανείς σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρώτες ύλε που ε, θα πρέπει να τις διαπραγματευτούμε σε σχέση με, με τις πρώτες ύλε που έχουμε στην Ευρώπη. Δύσκολες διαπραγματεύσεις και πρόκειται για πολλούς τομείς Υπάρχουν πρώτες ύλε που υπάρχουν, που είναι διαθέσιμες στην Ευρώπη, για τις οποίες όμως θα πρέπει να συνάψουμε νέες συμφωνίες. Έγιναν κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια για τα θέματα αυτά, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, γιατί σε, πολλής, σε πολλούς τομείς, όσον αφορά τις πρώτες ύλε, πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και η ανάπτυξή μας εξαιτίας της ελάχιστης πρόοδου που έχει γίνει. Χρειαζόμαστε επίσης και μια κοινή πολιτική δημιουργίας προτύπων, ιδιαίτερα με τους μεγάλους εμπορικούς μας εταίρους όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και με μεγάλες αναπτυσσόμενες αγοράς, αγορές στην Ασία, πάνω από ένα δισεκατομμύριο καταναλωτές, αγορές τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πιο δυναμικό τρόπο. Αποκινούμε τους Αμερικανούς. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το θέμα των κοινών προτύπων, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε επιτέλους να μιλήσουμε για διεθνή πρότυπα. Αυτές λοιπόν είναι οι γενικές μας στρατηγικές όσον αφορά τη δημιουργία ενός πλαισίου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος και βεβαίως αυτό είναι δύσκολο και μεγάλο έργο για εσάς κυρίες και κύριοι. Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο, τον κύριο Ρόιλ, και ξέρω ότι συμφωνεί μαζί μου ότι είναι απαραίτητο το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα του αντικτύπου της νομοθεσίας, του νομοθετικού έργου. Ποιες είναι οι οικονομικές, οι τεχνικές, οι κοινωνικές, οι οικολογικές συνέπειες μιας νομοθετικής πρότασης. Πολύ σημαντική πρόοδος έχει γίνει, όμως πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό και πιστεύω ότι στην νομοθετική του εργασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τον αντίκτυπο. Είναι κάτι που επαναλαμβάνω θα πρέπει να μας σας απασχολήσει ιδιαίτερα στο μέλλον. Όλα αυτά τα σημεία τα οποία σας παρουσίασα σαφώς και θα συμπεριληφθούν στην νέα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική ιδιαίτερα μετά την ε, κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας και η επόμενη Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειες για μια καλύτερη πολιτική στην Ευρώπη στον τομέα της απασχόλησης. Ξέρετε ποια είναι οι, ποιες είναι οι προτεραιότητες της Λισαβόνας για το θέμα της απασχόλησης και βεβαίως πιστεύω ότι το 2010 η συνάντηση κορυφής και το Συμβούλιο της Άνοιξης υπό Ισπανική Προεδρία θα δείξει ότι τα πρώτα καλά αποτελέσματα σίγουρα θα έχουν εμφανιστεί στην Ευρώπη. Αλλά σίγουρα μια καλύτερη εταιρική σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών δεν μπορεί παρά να βοηθήσει εδώ στην ανάκαμψη και στην υλοποίηση μιας νέας πολιτικής στον τομέα της βιομηχανίας και σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μία απρόσκοπτη, συνεκτική πολιτική με σκοπό να υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής, αύξηση της ανταγωνιστικότητας από τη μία και βιώσιμη ανάπτυξη από την άλλη. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πολιτικό απτό αποτέλεσμα, αν θέλετε, των τελευταίων ετών είναι ότι υπήρχε και υπάρχει ομοφωνία στην Επιτροπή η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη δεν θα πρέπει απλώς να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα από άποψης τεχνολογικής, αλλά και ιδιαίτερα να ληφθεί υπόψη η εξοικονόμηση της ενέργειας, η βιωσιμότητα και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η αντιπαράθεση μεταξύ οικονομίας και οικολογίας είναι κάτι το απαρχαιωμένο. Σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μεγάλα παγκόσμια προβλήματα, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται η αηφόρος ανάπτυξη, η βιωσιμότητα, η χρηστή κατανάλωση των πρώτων υλών, των πόρων και της ενέργειας. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες τομεακές ε, δραστηριότητες που βεβαίως είναι αρμοδιότητα άμεση αυτής της Επιτροπής, όπως παραδείγματος χάρη το παρατηρητήριο Global Monitoring Environment System, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη Γη. Το παρατηρητήριο αυτό έχει σαφώς προχωρήσει στη φάση της υλοποίησης. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τώρα την χρηματοδότησή του. Πρόκειται για ένα τεράστιο σχέδιο και θα πρέπει αφού διασφαλίσουμε τις πηγές χρηματοδότησης να σιγουρευτούμε ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. Να είναι γνωστές οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες σε όλους έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την υλοποίηση αυτού του σχεδίου στα πλαίσια των δαπανών και στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος. Περιμένουμε βεβαίως ακόμα. Πρόκειται όμως για κάτι που χρειάζεται μια σαφή απάντηση Υπάρχουν ε, εναλλακτικέ λύσεις με συγκεκριμένο κόστος. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο οικονομική λύση από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε ε, σφάλμα στην επιλογή μας. Το GMES είναι ένα σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι ένα κέντρο το οποίο θα αυτοχρηματοδοτείται από ένα σημείο και πέρα. Τώρα, το πακέτο φάρμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει τρία τμήματα, κάποια αμφισβητούνται και κάποια δεν αμφισβητούνται. αναφερόμαστε στα φάρμακα, στις απομιμήσεις φαρμάκων, στην ενημέρωση γύρω από τα φάρμακα αυτά και θα ήθελα εδώ να πω πολύ συγκεκριμένα ότι εγώ στηρίζω 100% αυτές τις προτάσεις και θεωρώ με πεπισμένος ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία οι πολίτες, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να καταλαβαίνουν τι συμπεριλαμβάνει ένα φάρμακο, να γνωρίζουν και ότι αυτές οι πληροφορίες δεν απευθύνονται μόνο σε φαρμακοποιούς και γιατρούς. Προς το παρόν είναι οι μόνοι που καταλαβαίνουν. Ο απλός άνθρωπος που θα πάρει το φάρμακο δεν καταλαβαίνει τι πληροφορίες του δίνονται. Παραδείγματο χάρη, είδαμε τι γίνεται με το εμβόλιο για την ε, γρήπη Α και τα υλικά τα οποία συμπεριλαμβάνει αυτό το εμβόλιο. Ξέρουμε σήμερα ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν δίνονται οι πληροφορίες όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό εξάλλου και οι γιατροί θέλουν να εμβολιαστούν. Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, λιγότερο ευχάριστο θέμα. Ξέραμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη βρίσκεται μπροστά από δύσκολες εποχές. Δεν πιστεύαμε ότι τόσο γρήγορα θα βυθιστεί στην κρίση. Εδώ υπάρχει βεβαίως συμφωνία όσον αφορά την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει αυτός ο βιομηχανικός τομέας και από τη μία υπάρχει σημαντική μείωση της ζήτησης, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν και οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες. Για πρώτη φορά ζούμε στον τομέα αυτό μία κατάσταση όπου όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν τα ίδια και σοβαρά προβλήματα. Την ίδια ώρα οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να αποφασίσουν πολύ σοβαρές επενδύσεις αν θέλουν να τηρήσουν τις ανώτατες ε, τιμές, τα ανώτατα όρια για τις εκπομπές ε, διοξιδιού. Είναι απαραίτητες αυτές οι επενδύσεις. Την ίδια ώρα όμως βεβαίως θα πρέπει να δούμε και την ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού. Επουδενή λόγο όμως δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Είναι δύσκολος ο δρόμος μέχρι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο. Και αν ε, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την αυτοκινητοβιομηχανία, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την μετάβαση από τον παραδοσιακό κινητήρα, τον σημερινό, στον κινητήρα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Καταλαβαίνετε ότι η μετάβαση δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει χωρίς πολύ σημαντικές ανακατατάξεις. Υπάρχει σήμερα πρόβλημα θέσεων απασχόλησης που θα καταστραφούν, που θα εξαλειφθούν και θα πρέπει εδώ και η Επιτροπή να λάβει το ρόλο της, τον ρυθμιστικό. Σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και κοιτάξτε τι γίνεται παραδείγματος χάρη σήμερα με την υπόθεση της General Motors και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων του ομίλου. Κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε ότι υπάρχει σήμερα μια κρίση η οποία έχει αντίκτυπο ετεροχρονισμένο. Εν πάση περιπτώσει, όλες οι χώρες που πλήττονται από το κλείσιμο αυτό του General Motors και την εξαγορά παίρνουν μέτρα για να αποδεσμευθούν από τον όμιλο, από την έδρα, από τη μητρική εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν κάποιες δυνατότητες επιβίωσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Και πρέπει να δώσουμε σε όλες τις τέτοιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη αυτή τη δυνατότητα. Και γι' αυτό το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και όλα τα κράτη-μέλη ε, δέχτηκαν την χρηματοδότηση όπως την είχε προτείνει η Γερμανία. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το είχαμε δεχτεί. Αλλά το κάναμε για να τους δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία. Και σήμερα πώς έχει η κατάσταση. Υπάρχει η τελική πρόταση για τη νέα εταιρεία και βεβαίως αυτή η νέα πρόταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά μόνο με κρατική υποστήριξη. Και βεβαίως το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα αυτές οι επιδοτήσεις πώς μπορούν να γίνουν δεκτές, υπό ποιους όρους και ποιες ε, προϋποθέσεις. Είναι δυνατό να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο, αλλά βεβαίως εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρήσει η Επιτροπή. Πρόκειται για επιδοτήσεις, πρόκειται για υποστήριξη, οι οποίες μπορεί να γίνουν ε, αποδεκτές παρά μόνο εάν το πρόγραμμα, το σχέδιο αυτό, το οποίο θα επιδοτηθεί, είναι οικονομικά βιώσιμο. Δεν μπορεί να είναι μόνο πολιτική η οι λόγοι για τους οποίους θα επιδοτηθεί ε, μία επιχείρηση. Δεν θέλω λοιπόν να προτρέξω της τελικής απόφασης. Η λύση είναι η καλύτερη. Ελπίζω να προχωρήσει αυτή η πρόταση και ελπίζω τουλάχιστον να μπορέσουμε να διατηρήσουμε α, τις επιχειρήσεις αυτές στην Ευρώπη που ανήκαν σε αυτόν τον όμιλο. Η Κομισιόν στηρίζει αυτή την προσπάθεια, αλλά βεβαίως θα πρέπει να τηρηθούν και κάποια κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις και επαναλαμβάνω το βασικό κριτήριο είναι να υπάρχει μια οικονομική βιωσιμότητα μακροπρόθεσμη. Αφού μιλάμε λοιπόν για οχήματα, δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα αυτοκίνητα, αλλά και για οτιδήποτε πετάει, επιπλέει. Αυτοκίνητα, αεροσκάφη και πλοία η κατάσταση είναι δραματική όσον αφορά παραδείγματος χάρη τα ναυπηγεία, μηδενική δραστηριότητα. Πριν από 15 μέρες οργανώσαμε ένα συνέδριο και όλοι οι συμμετέχοντες, οι περιφέρειες, ε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι επιχειρήσεις, και φτάσαμε σε κάποια συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις. Η Ευρώπη θα πρέπει να διατηρήσει κάποια ναυπηγεία. Θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Από την άλλη μεριά, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εξειδικευτούν αυτά τα ναυπηγεία. Δηλαδή να είναι εξειδικευμένα και τόσο υψηλής τεχνολογίας που να μην μπορεί κανείς άλλο στον κόσμο να τους ανταγωνιστεί. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί βιομηχανικοί τομείς έγιναν αντικείμενα σχεδιασμού έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Και αυτό το κάναμε βέβαια από κοινού με τα ενδιαφερόμενα κράτη, τις περιφέρειες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους ε, επιχειρηματίες, τις τοπικές αρχές και αναρωτιέμαι στο άμεσο μέλλον τι περιμένουν οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις από εμάς και τι περιμένουμε εμείς από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Εμείς καταρχήν καλούμεθα να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και όσον αφορά τη διαχείριση των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και όσον αφορά ε, τις επιπτώσεις και αυτό ισχύει για πολλούς τομείς όπως η χημεία, ε, η, ταναυπηγία η κλωστοεφαντουργία, η χαλιβουργία και τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών μέχρι τώρα στην Ευρώπη αποτελούν και τη βάση για τις προτάσεις της Επιτροπής που θα ενημερώνονται και θα δημοσιεύονται μετά βεβαίως και από ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο διαθετούμε μία μέθοδο δίκαιη, διαφανή, δημιουργώντας προϋποθέσεις και όρους για βιομηχανικούς τομείς, για αγορές, όπου όλα δεν είναι δημόσια και κρατικά, Ακούμε πολλές φορές κριτική όσον αφορά την μία ή την άλλη κατεύθυνση που παίρνει η ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά πραγματικά τίποτα δεν αποφασίζεται κρυφά με τους ε, επικεφαλής κάποιων επιχειρήσεων. Έχουμε μία μέθοδο ανοιχτής διαβούλευσης με διαφάνεια και με ανακοινώσεις και δημοσίευσεις. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε και αν υλοποιηθούν οι προτάσεις μιας τέτοιας διαβούλευσης να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά όσον αφορά την δημιουργία κάποιων προϋποθέσεων που θα πλαισιώσουν αυτήν την ε, πολιτική. Εγώ, ξέρετε, είμαι στο τέλος της πολιτικής μου θητείας και είναι, αν θέλετε, και η ώρα να κάνω και κάποιον απολογισμό. Θα ήθελα να σας αναφέρω ποια είναι αυτά που μου φαίνονται τα πιο σημαντικά. Για να διευκολύνουμε την ελευθερία των επιχειρήσεων και το πνεύμα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, θα πρέπει να απελευθερώσουμε τις επιχειρήσεις από υπερβολικά βάρη γραφειοκρατικά. Και δεν μιλάω για θέματα που είναι απαραίτητα, όπως η υγιεινή, ασφάλεια. Αναφέρομαι στο υπερβολικό βιογραφειοκρατικό άρθρο, το οποίο είναι άχρηστο και το οποίο αυξάνει και το κόστος της παραγωγής. Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεχίζεται. Πριν από λίγους μήνες προετοιμάσαμε και μια πολύ εντελεχή έκθεση όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει, διαβάζοντάς τη, ότι ο στόχος μας, ο οποίος έχει θυμάστε το 2012, που είναι η μείωση αυτού του γραφειοκρατικού άχθους κατά 25% έχει ως ένα βαθμό επιτευχθεί. 40 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που έχει μέχρι τώρα. Και βεβαίως εδώ θέλουμε και την βοήθεια του νομοθέτη, της νομοθετικής αρχής. Πρόκειται για τεράστια ποσά που μπορούν να εξοικονομηθούν εάν προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Είστε η Επιτροπή αυτή η οποία βεβαίως μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό και ζητώ ιδιαίτερα από σας την προσοχή σας για το σχέδιο αυτό. Τα τελευταία πέντε χρόνια, πρέπει να σας πω, χαρακτηρίζονται από θετικά και κάποια αρνητικά στοιχεία. Θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πολλές φορές ε, θέλει κίνητρα, περισσότερα κίνητρα. Η πολιτική παρέμβαση, η νομοθεσία θα πρέπει να είναι προσεκτική στο τι κάνει, στο τι αποφασίζει, έτσι ώστε να μην παρεμποδίσουμε την επιχειρηματικότητα. Και η άποψή μου είναι ότι η οικονομία της αγοράς με κοινωνική ευαισθησία θα πρέπει να επιτρέπει στους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν και ότι είναι μια πραγματική παρεξήγηση κατά την άποψή μου και πολλές φορές και οι πολιτικοί μου φίλοι κάνουν αυτό το λάθος. Μία πολιτική η οποία είναι φιλική προς τον επιχειρηματία δεν είναι απαραίτητα εχθρική προς τον εργαζόμενο. Αυτό είναι ένα σφάλμα που κάνουν πολλές φορές ε, πολιτικοί. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σαν πολιτικοί. Μπορούμε να διευκολύνουμε την κατάσταση. Αλλά η προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μία πολιτική η οποία να είναι φιλική προς τον επιχειρηματία, αυτό δεν σημαίνει επουδενή λόγο ότι τα συμφέροντα των επιχειρηματιών ξεπερνούν και επικρατούν επί των συμφερόντων των, της κοινωνίας. Δεν σημαίνει αυτό φιλική προς τον επιχειρηματία πολιτική. Σημαίνει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο προϋποθέσεων και συνθήκων έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να αναπτυχθούν, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Κάτι το οποίο είναι καθοριστικό για την εποχή που θα αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη από εδώ και πέρα. Θα πρέπει λοιπόν να κατευθύνουμε, να καθοδηγήσουμε την ε, αγορά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχουν συνεχώς νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτά ήθελα να σας πω Ξέρω ότι δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, δεν μπορώ εξάλλου. Βρισκόμαστε όμως στην αρχή μιας νέας ε, νομοθετικής περίοδου. Ήθελα λοιπόν να σας κάνω μια συνολική και γενική παρουσίαση αυτών που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό και αυτά που βρίσκονται ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτροπε για την πολύ λεπτομερή αυτή παρουσίαση που μας κάνετε και για το ειλικρινή κριτική και πλήρης σοφίας υποδείξεις τις οποίες μας κάνατε για να κάνουμε μια καλή εκτίμηση για τα προγράμματα με τα οποία θα ασχοληθούμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Και είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσουν βάση για συζήτηση και για κριτικές παρατηρήσεις και σχόλια. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ αγαπητοί συναδελφοί να είστε κάπως λακωνικοί. Γιατί όταν μιλάει κανείς δεν έχει την αίσθηση ότι ο χρόνος τρέχει. Θέλουμε όμως να μιλήσουν όσο πιο πολύ μπορούν. Για να έχουμε και απαντήσεις μετά, αν μην χρειαστεί να διακόψουμε βία. Η κυρία Δικαστήγιο πρώτη. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε εδώ σήμερα. Θέλω να επεφεληθώ μάλιστα από την ευκαιρία αυτή για να σας ευχαριστήσω για την δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα μαζί με τη δικιά μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή τα τελευταία πέντε χρόνια. Ήρθατε εδώ και έχετε αναλάβει την ευθύνη της βιομηχανίας και μαζί ε, συζητήσαμε πάρα πολύ γι' αυτά. Θέλω να επικεντρωθώ σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Τα Πρώτον, του χρόνου είναι το έτος καινοτομίας και δημιουργίας, το ευρωπαϊκό έτος δηλαδή καινοτομίας και δημιουργίας. Είναι η χρονιά που μάλιστα συμπίπτει με το τέλος ε, της ε, ατζέντα της Λισαβόνας. Η ατζέντα της Λισαβόνας, η στόχη της Λισαβόνας, όπως γνωρίζουμε όλοι, αφορά και την πολιτική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο ήταν ε, το πλαίσιο, το, το πλαίσιο αναφοράς επιμονή βάσεως, στο οποίο εμείς αφοσιώσαμε τις προσπάθειές μας. Προσπαθήσαμε δηλαδή να βοηθήσουμε για να δώσουμε και εμείς όθηση στις διάφορες αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη συζήτηση που γίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει τέτοια συζήτηση που γίνεται εδώ, στην οποία να μην αναφέρεται η ατζέντα της Λισαβόνας. Και όντως βοήθησε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι 10 χρόνια μετά εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα ανάμεσα, για παράδειγμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και μας. Δεν έχει μικρύνει αυτό το χάσμα σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας. Δυστυχώς το χάσμα αυτό έχει μεγαλώσει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω τον Επίτροπο γι' αυτό. Εσείς πώς βλέπετε την ανάπτυξη ενός σχεδίου πλαισίου, προς ποια κατεύθυνση, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει και να ανανεώσει τους στόχους της Λισαβόνας. Εγώ πιστεύω ότι η ανακοίνωση του Innovation Act που ε, Παρουσίαση Επιτροπή είναι κάτι σημαντικό και συμφωνώ με τα συμπεράσματα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θέματα όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία, η ευρωπαϊκή πατέντα, θέματα όπως οι επενδύσεις στην καινοτομία ή η συνεργασια τεχνολογία, επιχειρήσεις είναι πράγματα ζωτική σημασίας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε, εσείς πώς βλέπετε επ' αυτού τη δράση της Επιτροπής και θα μπορέσετε να πρικοδοτήσετε το πλαίσιο αυτό με ένα πλαίσιο αναφοράς το οποίο θα αποτελέσει τη συνέχεια κατά κάποιο τρόπο των στόχων της Λισαβόνας. Και κάτι άλλο συγκεκριμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να έχουν επιστώσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να έχουν κεφάλαιο στην τράπεζα. Είναι πράγματα που αποτελούν εμπόδιο προκειμένου να έχουν πρόσβαση με μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις πιστώσεις. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που μελετώνται αυτή την εποχή, αλλά ρωτάω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, σκοπεύει να κάνει κάτι κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας και τρίτον για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, πέρα από την περίπτωση της Όπελ. Εγώ σαν Ισπανίδα καταλαβαίνετε ότι θέλω να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στην ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής, αλλά νομίζω ότι εδώ υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Είναι σε διεθνές επίπεδο τι γίνεται με την ανταγωνιστικότητα, γιατί δυσκολίες όπως αυτές που έχει η Γεωργία σήμερα, κάποια στιγμή θα περάσουν και σε άλλους τομείς άλλου είδους παραγωγή, εκτός από τα γεωργικά προϊόντα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, θα έχουμε παραγωγή που θα μπαίνει εκτός από, έξω από την Ευρώπη στην Ευρώπη και θα δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα με αυτά που έχουμε στη γεωργία σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Επίτροπο Μιλήσατε για την αυτοκινητοβιομηχανία, μιλήσατε για τα ανώτατα όρια όσον αφορά τις εκπομπές αερίων. Παίξατε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Η Επιτροπή έδειξε πνεύμα συμβιβασμού και συνένεσης και θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω γιατί Μιλήσατε για τις ε, προϋποθέσεις, πλαίσιο που θέλετε να δημιουργήσετε. Βρισκόμαστε όμως σε μια οικονομική κρίση. Και μιλήσατε, και αυτή είναι και η ερώτησή μου, για το μέλλον, για τις μελλοντικές τεχνολογίες. Μιλήσατε για τεχνολογίες ε, με πολύ χαμηλό άνθρακα. Μιλήσατε επίσης για την αποθήκευση ενέργειας, είτε αυτή ε, θα χρησιμοποιηθεί σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είτε κάπου αλλού. Και εδώ ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Όλοι οι αυτοκινητοβιομηχανοί σήμερα παρουσιάζουν ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, συγγνώμη, τα οποία όμως έχουν πρόβλημα αυτονομίας. Έχουν πρόβλημα πώς θα αποθηκεύσουμε την ενέργεια και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις τεχνικές δυσκολίες. Σήμερα Ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στην ε, έρευνα, στην έρευνα που όπως ξέρετε επικεντρώνει τις ε, προσπάθειές της σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σχέδια, όπως παραδείγματος χάρη στο κινητό βιομηχανία, ενέργεια. Εσείς λοιπόν σαν Επιτροπή θα πρέπει να ασκήσετε περισσότερες πιέσεις όσον αφορά τις επενδύσεις και τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν σε αυτούς τους τομείς της έρευνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, επειδή μιλήσατε για τον αντίκτυπο της πολιτικής. Βεβαίως, η πολιτική έχει οικονομικό αντίκτυπο, κοινωνικό αντίκτυπο και κυρίως αντίκτυπο επί της απασχόλησης. Ζητούμε λοιπόν και εμείς από την πολιτική όταν αποφασίζεται μια στρατηγική και μια πολιτική κατεύθυνση και αν θέλουμε να φέρουμε τον Ευρωπαίο πολίτη κοντά μας και να δείξει εμπιστοσύνη, θα πρέπει να γίνεται αντίκτυπος και αξιολόγηση και της κοινωνικής πτυχής αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φανμπρέμπτ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον Επίτροπο που ήρθε εδώ και τόσο ανοιχτά μας μίλησε δεν είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του. Χαίρομαι που τον άκουσα σήμερα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε πολύ καλά να συνεργαστούμε στο μέλλον. Σε στηρίζουμε λοιπόν. Και γιατί, γιατί πιστεύετε πραγματικά στην βιομηχανική πολιτική. Πιστεύετε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή και δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτά που πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι εδώ σε αυτή την Επιτροπή πιστεύουμε ότι είναι. Δηλαδή ότι θέλουμε μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη με μια πολύ σημαντική ε, πτυχή που να είναι η καινοτομία. Αναφερθήκατε στην τεχνολογία, στην κατάρτιση. Υπάρχει κάτι για το οποίο όμως θέλω να σας ρωτήσω εγώ πολύ συγκεκριμένα. Σε τι βαθμό η Επιτροπή δουλεύει πάνω σε μια νέα ιδέα για τη βιομηχανία που έχει να κάνει με το from cradle to cradle, δηλαδή αυτό το οποίο ε, παράγεται να είναι εχμής, να είναι στο πιο ψηλό επίπεδο. κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα της βιομηχανίας μας. Και κάτι άλλο, και συγγνώμη τώρα γι' αυτό, είμαι βέβαια Βελγίδα, στην Αβέρσα ζω και θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα για την Όπελ στην Αβέρσα. Ήσασταν ανοιχτό απέναντί μας και συμφωνώ με αυτά που είπατε εσείς, ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν συμφωνούν με αυτά τα οποία σήμερα συμβαίνουν. Διαβάστε τις εφημερίδες να δείτε τι λένε. Εσείς μας είπατε ότι οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν μόνο εφόσον βασίζονται σε οικονομικά επιχειρήματα. Συμφωνώ, αλλά τα οικονομικά επιχειρήματα πούντα. Με άλλα λόγια, εμείς και όχι μόνο η βελγική, η φλαμανδική κυβέρνηση δεν βλέπουν αυτά τα οικονομικά κριτήρια που σήμερα καθορίζουν την τύχη της Όπελ. Που λειτουργεί πολύ καλά και είναι αποτελεσματική. Τη Δευτέρα λοιπόν διάβασα στον ε, τύπο, αλλά φαντάζομαι και στο Σπίγκελ θα το διαβάσατε, που αναφέρεται στην Όπελ. Λέει η γερμανική κυβέρνηση ότι βάσει αυτών των οικονομικών κριτηρίων το εργοστάσιο στην Αμβέρσα είναι λιγότερο αποδοτικό από ό,τι εκείνο στον Πόχουμ. Ρωτάω λοιπόν, αυτό το αποφασίζει η γερμανική κυβέρνηση. Μπορεί να καθίσει αυτό να το γράψει και να το δώσει στον τύπο. Να υπάρξει τέτοια διαρροή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους στην Αβέρσα να τους λέτε ότι δεν είναι αποδοτική. Και ποια είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θα κάνει η Επιτροπή. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τελικά αυτά τα οικονομικά κριτήρια. Πότε θα πει κάτι συγκεκριμένο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα το κάνει όταν θα είναι πια πολύ αργά. Με άλλα λόγια, επειδή μιλάμε ειλικρινά μεταξύ μας, θα ήθελα να ξανανοίξετε τον τοσχέτη της Όπελ. Έχω την εντύπωση ότι το μόνο που πραγματικά ευρωπαϊκά δουλεύει σήμερα είναι τα συνδικάτα. Μόνο τα συνδικάτα σήμερα τολμάνε να μιλάνε για αλληλεγγύη. Κάτι για το οποίο εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή δεν μιλάει αρκετά. Γιατί καλά όταν πάνε ωραία τα πράγματα, αλλά και όταν δεν πηγαίνουν καλά, πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη μεταξύ μα. Ευχαριστώ να μου απαντήσετε στην ερώτησή μου. Ο κύριο Γκέρεκ. Dziękuję Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, παράγεται με αυτό που ανάφερε πριν η συνάδελφος για την Όπελ. ήταν το κέντρο της παρέμβασής της η ΟΠΕΛ. Εγώ έχω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Παραμένω στο θέμα ΟΠΕΛ. Ο καναδικο-ρωσικός όμιλος δεν μπορεί να δημιουργήσει μετατόπιση του εργοστασίου έξω από τα σύνδρα της Ένωσης. Στην Πολωνία ήδη συζητιέται να φύγει το εργοστάσιο από το Κλίβιτς και να πάει στη Ρωσία. Αληθεύουν αυτά. Τι ασφάλεια έχουμε εκ μέρους της Κομισιόν ως προς ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί αν ήταν απλώς θέμα ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας, με την κατάσταση προς τη Ρωσία, ίσως να εμπερίχει ένα στοιχείο ανταγωνισμού, γιατί εκεί δεν συζητάνε για τα εργατικά στη Ρωσία, δεν συζητάμε. Η ποιότητα όμως είναι άλλο θέμα. Η ποιότητα θα είναι χειρότερη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίτης. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti gerbiamam komisarui už Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και εγώ για τη τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Μας μίλησε για τις προπτικές της βιομηχανίας μας. Εγώ είμαι καινούριο ευρωβουλευτής. Όμως, εκπροσωπώντας τη χώρα μου, θέλω και εγώ να θέσω σοβαρά ερωτήματα. Βρισκόμαστε μέσα σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Η Επιτροπή λοιπόν μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέτος έκανε μια έρευνα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έρευνα αφορά και τις 27 χώρες, αλλά κυρίως την Ευρωζώνη επικεντρώνεται. Πολλές επιχειρήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζουν προβλήματα με χρηματοδότηση πήραν χρήματα από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από άλλα ταμεία. Άλλες χώρες μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες με τη χρηματοδότηση. Κύριε Πίτροπε, ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη στο μέλλον δεν θα έπρεπε να διατίθεται προς όλα τα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό στο οποίο αναφερθήκατε εσείς νωρίτερα, δηλαδή να πετύχουμε το στόχο της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και όλες τις άλλες πτυχές, δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Αυτή είναι η ερώτησή μου για να έχουμε ανταγωνιστικότητα και αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Eh, η κυρία Καβαλίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ που ήρθατε και μας δώσατε αυτές τις εξηγήσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό που η Επιτροπή αντιμετωπίζει οριζόντια την καινοτομία. Έχουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις μπροστά μας ως Ευρώπη και απαιτούνται συνολικές σφαιρικές απαντήσεις. Η πολιτική κοινοτομίας λοιπόν, κοινοτομίας, θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο και των άλλων πολιτικών, όπως μας είπε και ο Επίτροπος εξάλλου. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να σας ρωτήσω τώρα κύριε Επίτροπε, Συγκεκριμένα, πώς βλέπετε εσείς αυτή την στρατηγική υπέρ της καινοτομίας, πώς θα βοηθήσετε για τις τεχνολογικές αλλαγές που πρέπει να λάβουν χώρα. Είτε πρόκειται για μεταφορές, είτε πρόκειται για ε, ναυτιλία, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο. Είναι πολλοί τομείς βιομηχανικοί που καταναλώνουν ενέργεια και αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτία του περιορισμού εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είτε πρόκειται για την κεραμική, είτε πρόκειται για άλλους τομείς. Χρειάζεται συνέχεια μεταφορά τεχνολογίας. Η πολιτική καινοτομίας λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρότεινε η Επιτροπή, αυτή η πολιτική πώς θα βοηθήσει στις ε, μετατροπές που χρειάζονται. Ευχαριστούμε ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας μαζί μας. Ξεκίνησα με τα γερμανικά, συνεχίζουμε με τα ολλανδικά, ξέρω ότι τα καταλαβαίνετε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σας, όποια και αν είναι αυτή. Για την αυτοκίνητο βιομηχανία, Επίτροπε, ακούσαμε πολύ κριτική δεν αναφέρεται σε εσά απαραίτητα, σε όλη την Επιτροπή για την αντιμετώπιση που είχε η Επιτροπή απέναντι στην αταβιομηχανία τον τελευταίο καιρό. Θυμόμαστε από το 80 που είχαμε την κρίση του Χάλιβα. Ε, τα θυμίζει αυτά η σημερινή κρίση. Ξέρετε, η συνθήκη του Χάλιβα έχει αντικατασταθεί βέβαια. Κι άλλοι αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι θα έπρεπε εμείς να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να προλαβαίνουμε τα γεγονότα και όχι να δρούμε όταν είναι πολύ αργά. Και δεν πρέπει να υπάρχει εθνικισμός, να αρχίσουν να λέει «Μάμα, γιατί η Γερμανία έδωσε αυτά, γιατί η Αγγλία έδωσε αυτά, γιατί η Ισπανία έδωσε τα άλλα». Αν μπούμε σε αυτά δεν κερδίζουμε τίποτα, πρέπει να τα αποφεύγουμε. Συντονισμός χρειάζεται και υπάρχουν περιθώρια για συντονισμό σήμερα. Πιστεύω ότι και το προσπαθήσαμε λίγο πολύ, αν και είναι αμφίβολα τα αποτελέσματα, οι μεγάλοι παίκτε σε αυτό το τομέα να συνεχίσουν να μιλάνε, να συνεχίσουν να συζητάνε για την τεχνολογία και να συντονίζουν τη στρατηγική. Λέτε ότι είμαστε στο πιο χαμηλό σημείο της κρίσης και ότι θα αρχίσει η ανάκαμψη. Υπάρχουν διακυμάνσεις βέβαια. Η νέα γενιά οχημάτων λένε ότι θα είναι το ηλεκτρικό, αν και δεν είναι για μεθαύριο. Ναι, αλλά κάπου υπάρχει, είναι περίπου έτοιμο. Η αγορά λοιπόν, ίσως όταν δει τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να τα βοηθήσει να προχωρήσουν πολύ. Αλλά μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Αν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες ε, διώξουν προσωπικό. Αυτό πρέπει να δούμε. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Και εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα άρθρο στην Βίρτσες Βόχα. Χτες νομίζω ήτανε. Αναφέρθηκε κάποιος συνάδελφος αυτό. Αναφέρεται σε μια πολωνική εταιρεία η οποία μετεκαθίσταται στη Ρωσία. Είναι το ίδιο όπως και η ιστορία με την Αμβέρσα που φεύγει η επιχείρηση από εκεί και πάει στη Ρωσία. Εδώ νομίζω ότι μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί όταν υπάρχει στήριξη από την Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρχει μια προϋπόθεση, να μην υπάρχει τέτοια μετεκατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να στηρίζει η Ευρώπη και μετά να φεύγει η τεχνολογία αυτή και να πηγαίνει στη Ρωσία. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να παρέμβουμε. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα στην αυτοκινητοβιομηχανία ότι αν θέλετε να σας βοηθήσουμε στην τεχνολογία θα μείνει στην Ευρώπη. Και δεν θα φεύγει να πάει στη Ρωσία. Οπότε τελικά το ζήτημα είναι να μην μένει σε θελοντική βάση αυτό, αλλά να υπάρχει κάποια δέσμευση. Ευχαριστώ. Ähm, Σας ευχαριστώ. Έχω ακόμα έξι ομιλητές στον κατάλογο. Αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε σύντομα, κύριε Επίτροπε, γιατί αλλιώ θα είναι ακόμα πιο περίπλοκο για τους συναδέλφους. Πρέπει στις 4.30 να σας απελευθερώσουμε γιατί έχουμε καλέσει κάποιον άλλον. Ναι, θα προσπαθήσω όλες τις ερωτήσεις που έχουν σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία να τις συγκεντρώσω. Κυρία Καστήλο πέρα. σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε. Δεν είναι τόσο αρνητικά αυτά τα φαινόμενα. Ιδιαίτερα αν τα συγκρίνει κανείς με την παραγωγικότητα, τη δυνατότητα για καινοτομία, η θέση μας σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και με άλλους οικονομικούς χώρους στον κόσμο έχουμε βελτιωθεί. Δεν είναι βέβαια αρκετή η βελτίωση. Και η νέα ατζέντα, δηλαδή από αυτήν που καθορίσαμε το 2002 στη Λισαβόνη και την ενημέρωσή της το 2004 μας έχει οδηγήσει στο νέο πρόγραμμα που επεξεργαζόμαστε. Εμείς βασιζόμαστε σαφέστατα σήμερα σε στοιχεία του 2005 με μια νέα, αν θέλετε, ατζέντα της Λισαβόνας, άλλη από αυτή του 2000 βέβαια, διαφορετική, και με κάποιους στόχους που ενδεχομένως αμφισβητούνται πλέον το 2010 με την σημερινή κατάσταση. Δεν ξέρω πότε θα πετύχουμε και θα λεωποιήσουμε αυτούς τους στόχους έτσι όπως τους είχαμε θέσει τότε. Εν πάση περιπτώσει, η επόμενη θητεία, η επόμενη πενταετία αν θέλετε, σαφώς και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα και την εμπειρία των τελευταίων ετών έτσι ώστε να βελτιωθεί το σχέδιο το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε διατήρηση θέσεων απασχόλησης, δημιουργία νέων και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η πολιτική μας στον τομέα της ανάπτυξης μας έχει βοηθήσει. Η εμπειρία είναι καλή και σήμερα έχουμε μηχανισμούς στη διάθεσή μας που μας επιτρέπουν να ξαναχρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία που έχουμε. Υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα αμοιβαία ενημέρωσης, ανταλλαγής διδαγμάτων, και εμπειριών στην Ευρώπη. Η δυνατότητα λοιπόν για νέες τεχνολογίες, για καινοτομία, η ανταγωνιστικότητά μας, αν συγκριθεί με άλλα μέρη στον κόσμο, είμαστε στην πιο σημαντική ομάδα. Όσον αφορά την, την καινοτομία, παραδείγματο χάρη, η Ελβετία βρίσκεται με τη Φιλανδία και τη Σουηδία στην πρώτη γραμμή και ακολουθούν οι Αμερικανοί. Σε όλους τους τομείς λοιπόν βλέπετε ότι στην ομάδα κορυφής υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούμε λοιπόν να το καταφέρουμε, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και αυτό η αμοιβαία, αν θέλετε, ενημέρωση, γνώση, η μεταφορά ε, νέων τεχνολογιών, εμπειριών από τη μία χώρα στην άλλη μας έχει οδηγήσει σε αυτό το τόσο θετικό αποτέλεσμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βέβαια, οι συμφωνίες για τις εμπορικές συναλλαγές. Ναι. Δεν μίλησα πολύ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είναι, αν θέλετε, πολιτικό το πλαίσιο το οποίο δημιουργήσαμε. Και βρισκόμαστε στη φάση της υλοποίησης Τώρα, η πολιτική δανειοδότησης και χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ξέρετε, διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Υπάρχουν κράτη με μεγάλες τράπεζες, η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Άλλες χώρες με άλλο τραπεζικό σύστημα, διαφορετικής μορφής, με συνεταιριστικές τράπεζες, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα στηρίζονται περισσότερο οι μικρομεθαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τώρα έχει κάποιες δυνατότητες, αλλά αν κοιτάξει κανείς τα ποσά των διατραπεζικών δανείων στην Ευρώπη, πολύ περισσότερη ε, προσπάθεια χρειάζεται. Ο κύριος Γκρότε έκανε μια ερώτηση για την αυτοκινητοβιομηχανία, την αξιολόγηση του αντικτύπου του κοινωνικού. αυτό είναι προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βεβαίως, ε, αν υπάρχει και πίεση του Κοινοβουλίου, αυτό θα είναι πάντα πολύ χρήσιμο. Ναι, άλλη μια ερώτηση για την Όπελ. Κύριος Γκέρεκ επίσης. Ο κύριος Μπαλατσίτης. Μίλησα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι σωστό ότι μόνο στην Ευρωζώνη υπάρχει στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να κάνει διάκριση αν είναι στην Ευρωζώνη ή όχι. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία είναι στην δική μου διεύθυνση και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου και αν βρίσκονται. Επίσης αναφερθήκατε στα δικαιώματα και στην στήριξη ή στήριξη για όλους. Αυτό δεν υπάρχει σαν έννοια. Οι πιο αδύναμοι στηρίζονται περισσότερο. Οι ισχυροί δεν ενισχύονται. Η αρχή της αλληλεγγύης επικρατεί εδώ. Με σκοπό να εξισορροπηθούν οι ανισορροπίες που υπάρχουν. Αυτό είναι ο στόχος αυτής της πολιτικής. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που είναι καθυστερημένοι ακόμα. Αλληλεγγύη, λοιπόν, είναι μία από τις βασικές έννοιες της ευρωπαϊκής πολιτικής. κυρία Καβάλιο, συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες που μπορούν υπό τη μορφή εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να δώσουν όθηση σε κάποια από τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε. Βεβαίως και εδώ θα πρέπει να αποφευθούν οι επικαλύψεις και να έχουμε ταχύτατα αποτελέσματα. Υπάρχουν και άλλα πολιτικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να δώσουμε κίνητρα για την ε, τεχνολογική καινοτομία. Ρυθμίσεις, κανονισμοί, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τα ανώτατα όρια εκπομπών. Ναι, Σίγουρα αυτό μπορεί να δώσει μια επιπλέον όθηση και κίνητρα στην αυτοκινητοβιομηχανία για να αναπτύξουν τις καθαρές τεχνολογίες και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς. Το ερώτημα είναι πώς θα κατανείμουμε το βάρος όλων αυτών των διευθετήσεων που απορρέουν από το σύστημα εμπορίας των εκπομπών. Πώς θα γίνει η κατανομή των βαρών και τι θα κάνουμε με τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες καταναλώνουν πολλή ενέργεια και βεβαίως έχουν υψηλά επίπεδα εκπομπών, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής μας και δεν έχει νόημα εδώ αν αυτές οι επιχειρήσεις ε, πάψουν να είναι ανταγωνιστικές και τα ίδια προϊόντα συνεχίζουν να παράγονται παλού στο, παντού στον κόσμο. Όλοι οι τομείς και υποτομής της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής αναλύονται της ευρωπαϊκής οικονομίας από την Επιτροπή. Και βεβαίως όσον αφορά την διαρροή του άνθρακα, το carbon leakage, άσχετα με το ποιες είναι οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, θα πρέπει να ειδωθούν υπό το πρίσμα των οικολογικών επιπτώσεων, της μόλυνσης που προκαλούν. Και πιστεύω ότι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν σε σημαντική τεχνολογική πρόοδο. Τώρα, όσον αφορά τα αυτοκίνητα. Σε γενικές γραμμές όσον αφορά το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Εγώ θεωρώ ότι όταν ξεκινήσαμε με τα πρώτα μέτρα το 2004, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι στην Ευρώπη έχουμε το πιο σύγχρονο μοντέλο πρότυπο αυτοκινητό βιομηχανία στον κόσμο. Και θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, η κρίση είναι κάτι που δεν οφείλεται σε αιτίες βιομηχανικής πολιτικής. Η Επιτροπή θέλει να θέσει συγκεκριμένα κίνητρα και όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, το σύστημα των επιδοτήσεων, των κινήτρων, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη ανάλυση. Δεν είναι δυνατόν η Επιτροπή να δώσει ούτε ένα ευρώ για μη βιώσιμα μοντέλα. Και οι επιδοτήσεις στο ευρωπαϊκό ε, δίκαιο, αν θέλετε, απαγορεύονται. Αν διαβάσει κανείς τις συνθήκες, βλέπει ότι απαγορεύονται. Απλώς υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπου επιτρέπονται. Και μπορεί η Επιτροπή σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει αυτές τις επιδοτήσεις και με πολύ συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Από τα διαρθρωτικά ταμεία μπορεί να δοθούν κάποια ποσά για στήριξη των επενδύσεων. Αυτό όμως υπό όρους και προϋποθέσεις επαναλαμβάνω είναι παράλογο να στηρίξουμε παραδείγματο χάρη μια επιχείρηση επιδοτώντας τις επενδύσεις τους χωρίς αυτοί να έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης παραδείγματο χάρη. Όσον αφορά την κρατική παρέμβαση σε μια αγορά, αν μια επιχείρηση ή ένας τομέας ολόκληρος είναι σε δυσκολία, εκεί μπορεί εξαιρετικά να επιτραπεί η ενα τομεα ολοκληρο ειναι σε δυσκολια εκει μπορει εξαιρετικα να επιτραπει η επιδοτηση και από την πρώτη ημέρα αυτής της ε, συζήτησης ήμασταν σαφέστατοι. Είπαμε θα επιτραπεί αυτή η στήριξη μόνο και εφόσον υπάρχει ένα συγκεκριμένο business plan, ένα σχέδιο επιχειρησιακό, το οποίο να δείχνει ότι υπάρχει βιωσιμότητα οικονομική και επιπτώσεις θετικές στην αγορά εργασίας. Η Επιτροπή λοιπόν διασφάλισε σε τρεις υπουργικές, αν θέλετε, συναντήσεις και με μια τεράστια, αν θέλετε, προσπάθεια συνεδριάσεων και συναντήσεων και παρουσία και της βελγικής και της φλαμανδικής κυβέρνησης. Και δεν είναι αλήθεια ότι έγινε ερήμην της βελγικής κυβέρνησης αυτή η απόφαση. Όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις γνωρίζουν το τελικό σχέδιο, το οποίο μας έχει υποβάλει η επιχείρηση και η Ισπανική και η Πολωνική και η Βρετανική κυβέρνηση γνωρίζουν το σχέδιο αυτό, έχουν ενημερωθεί και η προθεσμία είναι μέχρι αύριο. Και κατόπιν όλοι μπορούν να αποφασίσουν, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν ναι ή όχι θα δοθούν βοήθειες και τελικά η Επιτροπή έχει πει με μεγάλη σαφήνεια ότι θα ελέγξει όλες τις επιδοτήσεις που ενδεχομένως θα δοθούν και ότι ε, που δεν είναι λόγο δεν θα πρέπει να δοθούν επιδοτήσεις σε καθαρά πολιτικούς ε, προσανατολισμούς. Δεν θα του δεχτούμε. Χρειάζεται ένα οικονομικά βιώσιμο πλάνο. Τώρα, όσον αφορά την ποιότητα αυτών των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ευρώπη, η γερμανική κυβέρνηση μα δεν έχει ούτε τη δυνατότητα, ούτε την ιδιότητα να κάνει μια τέτοια αξιολόγηση της ποιότητας. Αυτό μπορεί να το κάνει ο παρόν και ο μέλλον ιδιοκτήτης. Δεν ξέρω τι είπε η γερμανική κυβέρνηση. Αν είπε κάτι, σίγουρα βασίστηκε σε στοιχεία του παλαιού ή του νέου ιδιοκτήτη. Μπορούμε, αν θέλετε, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν κάποιες ε, πληροφορίες που είναι απόρριτες για το θέμα αυτό. Αλλά ο παλιός ιδιοκτήτης της επιχείρησης σίγουρα κάνει τελείως διαφορετική αξιολόγηση από τον καινούριο. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ της αξιολόγησης του ενός και του άλλου. Και εγώ πιστεύω ότι το εργοστάσιο στην Αμβέρσα έχει ελπίδες επιβίωσης και ότι πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά θα σας πω και κάποια άλλα πράγματα αργότερα, κατηδίαν. Μεταφορά τεχνολογίας προς τη Ρωσία. Αυτή η μεταφορά τεχνολογίας γίνεται καθημερινά. Καθημερινά μεταφέρουμε τεχνολογία στην Κίνα και σε άλλε χώρε. Το θέμα είναι πώς γίνεται, ποιε είναι οι προποθέσει αυτή τη μεταφορά τεχνολογίας. Ανήκουμε σε μια κοινωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει αυτήν την μεταφορά τεχνολογίας, είτε στη Ρωσία είτε αλλού. Και αυτό χωρίς άδειες, χωρίς παρατήρηση των ε, κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τις μεταφορές και με την καταστάσεις εργοστασίων, κατά την άποψή μου, η General Motors πήρε μια τέτοια απόφαση σχεδιάζοντας να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της Opel στην Ευρώπη καθώς και τις δυνατότητες παραγωγής στη Ρωσία και να δημιουργήσει εκεί ένα νέο πρότυπο αυτοκινήτου που να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στη ρωσική αγορά. Τώρα, αν οι Ρώσοι αργότερα γίνουν τόσο παραγωγικοί που μπορούν να εξάγουν στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Κινέζοι εξάλλου, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό πάντως που σήμερα προβλέπετε είναι να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο για τους Ρώσους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά κάτι το εξαιρετικό. Είναι μια τρομερή ευκαιρία για την Ευρώπη. Τελειώνοντας για τις μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων, δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς κυρίες και κύριοι. Μια επιχείρηση επιλέγει τον τόπο εγκατάστασής της βάσει κάποιων κριτηριών. Αν ο μόνος, ε, το μόνο κριτήριο είναι το κόστος των μισθών του προσωπικού, των εργαζομένων, δεν πρόκειται ποτέ μια εταιρεία να παραμείνει εκεί που έχει εγκατασταθεί. Ήταν στη Λιθουανία και θα φύγει εκτός Ευρώπης. Δηλαδή είναι ψευδέστηση και αυταπάτη αν μια επιχείρηση που διαλέγει αυτό το κριτήριο και θεωρεί ότι μπορεί να παραμείνει στην Ευρώπη. Εάν ξεκινήσει η προσπάθεια μείωσης των μισθών, τότε η Ευρώπη δεν θα κρατήσει καμία επιχείρηση. Δεν μπορούμε στην Ευρώπη να πληρώνουμε όλο και χαμηλότερους μισθούς. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν μπορεί να είναι στο πιο χαμηλό επίπεδο μιας αλυσίδας κόστους. Είμαστε στο πιο ψηλό σκαλοπάτι και θα πρέπει να είμαστε σε έναν ανταγωνισμό όσον αφορά την τεχνολογία και όχι όσον αφορά το κόστος των μισθών. Και για να σας μιλήσω πάλι για το θέμα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ένα μεσαίο αυτοκίνητο έχει μειώσει την τιμή του τα τελευταία χρόνια. 45.000 ευρώ. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό της μισθοδοσίας. 1.300 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και για πολύ ακριβά αυτοκίνητα είναι περιθωριακό το κόστος αυτό. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη έχει μέλλον. Δυστυχώ δεν τήρησα το χρόνο που είχα στη μου κύριε Πρόεδρε, αλλά νομίζω ήταν πολύ σημαντικές οι απαντήσεις. Έχετε δίκιο. Και ο χρόνος όμως είναι πολύ σημαντικός. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ζητήσουμε τον επόμενο επισκέπτη μας να περιμένει λίγο. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές και όλοι να είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Έχω μια ολόκληρη σειρά, επτά ομιλητές. Ο συνάδελφο, ο κύριος Μπίτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, κύριε Φερχόγεν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μας κάνατε. Λυπούμε, γιατί τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα είστε στην πρωτοπορία αυτών των αγώνων και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει μέλλον όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας και ότι πραγματικά πρέπει να δούμε και το θέμα της αηφόρου ανάπτυξης, της βιωσιμότητας αυτών των βιομηχανικών σχεδίων και θεωρώ ότι αυτά τα δύο κριτήρια τα αποφασίζουν σχεδόν όλα. Εάν Θέλουμε να υπάρξει πολιτική στήριξη για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, η οποία να έχει μέλλον. Χρειαζόμαστε κατά κάποιο τρόπο μια ιστορία, μια κεντρική ιδέα, η οποία να μπορέσει να εμπνεύσει και να βασίζεται σε μια οικολογική βιομηχανική επανάσταση. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε και να το ενισχύσουμε σαν μήνυμα, γιατί εδώ διαβάζοντα τον τίτλο όσον αφορά το carbon leakage, κατά κάποιο τρόπο συμπεριλαμβάνεται σε όλους τους τομείς της βιομηχανικής δραστηριότητας και προβλέπονται χιλιάδες εξαιρέσεις. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η καινοτομία θα πρέπει να επικεντρωθεί ακριβώς αυτούς τους τομείς. Δεύτερον, πιστεύω ότι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην πρωτοπορία. Με το πλάνο Ομπάμα 2,3 δις επενδύονται στην ε, ηλεκτρονική πρόθεση αυτοκινήτων. Οι Κινέζοι 75. Καταλαβαίνετε ότι εδώ χρειάζεται τεχνολογικό άλμα και δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είμαστε τοποθετημένοι σωστά στον τομέα αυτό. Και μια τρίτη παρατήρηση. Έχετε δίκιο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά μας σε σχέση με τους υπερατλαντικούς μας ε, συμμάχους. Θα ήθελα, κύριε Φερχόγγεν, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και εμείς, να δώσουμε περισσότερη σημασία στη συνεργασία μας με τις ε, χώρες τις λιγότερο αναπτυγμένες. Ευρωπαϊκή και Κινέζικη συνεργασία. Νομίζω ότι οι προσπάθειές μας για την εξάλληψη των δασμών θα πρέπει να είναι εξίσου σημαντική με αυτή που κάνουμε για τη δημιουργία των κοινών προτύπων όταν διαπραγματευόμαστε με τους Αμερικανούς. Τέλος, μιλήσατε για την στήριξη και είπατε ότι οι επιδοτήσεις θα δίνονται μόνο και εφόσον υπάρχει οικονομικό βιώσιμο μοντέλο. Δεν απαντήσατε όμως την ερώτηση για τον Όμιλο Μάγνα. Σας φαίνεται λογικό το σχέδιο αυτό. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για στήριξη και επιδότηση απαραίτητων καινοτομιών και τεχνολογικών αλμάτων, που είναι απαραίτητες και όχι στην επιδότηση παρχαιωμένων μοντέλων. Λόγω σας να Μπενότσινα και σας παρακολούμε να είστε λακωνικοί όλοι σας. Øh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Άκουσα με πάρα πολύ ευχαρίστηση τις παρατηρήσεις σας για το ότι δεν πρέπει να προωθεί προστατευτική βιομηχανική πολιτική. Επίσης, ο Επίτροπος μας είπε ότι η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη σιγά σιγά προχωράει μετά τα προβλήματα του 2008 και το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να προέρθει και από τα προγράμματα βοηθείας των εθνικών κυβερνήσεων. Η ερώτηση μου όμως κύριε Επίτροπε Φερχόγγιν είναι η εξής. Συμφωνείτε με το ότι πέρασε ο καιρός των ενισχύσεων και τα χρήματα του φορολογούμενου πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση, την καινοτομία, την έρευνα για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας και όχι να χρησιμοποιείται για υποστήριξη βιομηχανιών οι οποίοι δεν αντέχουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Γιατί έτσι θα χαθούν θέσει απασχόληση. Πρέπει χάρη τα περισσότερα ναυπηγεία στη Δανία αποφάσισαν να κλείσουν. Στη Γερμανία, στη Βαλτική το ίδιο. Στη Δανία στοιχίζει 25 εκατομμύρια δολάρια επιπρέον να φτιάξουμε ένα δεξαμενόπλιο, ένα κοντέινερ στη Δανία, στην Ευρώπη, από ό,τι στοιχίζει στην Ασία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για την καινοτομία ή για κρατικές επιδοτήσεις. Κατ' Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για καινοτομία, για την ανάπτυξη, για να καταρτήσουμε, να αυξήσουμε τις δεξιότητες των εργαζομένων μας. Δεύτερη ερώτηση. Έχουμε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πού είναι η ραχοκακαλιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Άκουσα τις παρατηρήσεις σας για, την, για τις διάφορες συμφωνίες. Το ερώτημα είναι οι όροι ανταγωνισμού, αυτό που λέτε level playing field, οι ίσοι όροι παιχνιδιού για όλους, θα ισχύσουν χωρίς να υπάρχει πρόσβαση και για μας στην αγορά των άλλων, όπως οι άλλοι έχουν πρόσβαση στην αγορά μας. Αυτό είναι αποφασιστικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στις εξωτερικές αγορές στο μέλλον. Όσο θα αυξάνει η αγοραστική δύναμη, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν προβλήματα με τις συμφωνίες τους και με τη θέση απασχόληση προσφέρουν αυτές. Οι συμφωνίες λοιπόν ελευθέρω εμπορίο, ιδιαίτερα όσον αφορά την τελευταία με την Κορέα, ξεκινά από την υπόθεση ότι κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστούμε επόμενο συνάδελφος. Ο κύριος Μπάλτσο, κύριε Επίτροπε, δεν είναι σύμπτωση το ότι πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δέστε τι γίνεται με τις τράπεζες. Σιγά αλλά σταθερά ξανασηκώνεται και στείνεται στα πόδια του. Βέβαια, αφιερώσετε αρκετό χρόνο γι' αυτό και σχεδόν μία πρωτοσούλα μόνο είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο μεγάλος χαμένος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάμε για πακέτα που βοηθούν να μην χρεοκοπήσουν επιχειρήσεις. Καλό είναι αυτό. Αλλά είναι σωστό να χρησιμοποιούμε και να στηριζόμαστε μηχανισμούς που επιτρέπουν την αυτορύθμιση των αγορών. Θα πρέπει να δούμε και ένα άλλο σενάριο. Ο περιορισμός των πιστώσεων έχει επίπτωση στις επιχειρήσεις, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στην Αμερική. Καλά είναι, καλός είναι ο ανταγωνισμός, αλλά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα ότι είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό κεφάλαιο το οποίο να διατίθεται στις επιχειρήσεις μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια από τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι το ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν καλύπτονται, οι πολυεθνικές καλύπτονται με κρατικές επιδοτήσεις για να μην χρεοκοπήσουν. Σωστό αυτό, διότι αν κλείσει μια τέτοια επιχείρηση θα έχουμε τεράστια απώλεια θέσεων εργασίας. Αλλά όταν μιλάμε για ασφάλεια, παραδείγματο χάρη ε, στην αεροναυπηγική κλπ., παρόλο ότι συμβαίνουν πολλά ατυχήματα και συμβαίνει ένα ατύχημα, μπορεί να σκοτωθούν χιλιάδε άτομα. Στατιστικά όμω, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί που σημειώνεται η ζημιά, η οικονομική ζημιά. Στη δική μας Επιτροπή ήδη γνωμοδοτήσαμε για τον προπολογισμό και λέμε να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίοι. Αυτό ισχύει, παραδείγματος πρέπει να ισχύει μάλλον και για την διασφάλιση τραπεζικών δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι η ραχοκοκαλιά της Ένωσης. Μιλάμε για ένα χρηματοπιστωτικό τσουνάμι, αν θέλετε. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν οι σωστές συνθήκες και ξέρω ότι αν τα δούμε τα πράγματα δογματικά όσον αφορά την ρύθμιση των χρηματαγορών, μπορεί να μην πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι μιλάμε για εξαιρέσει. Αλλά όλα αυτά είναι σε βάρος στις περισσότερες περιπτώσεις των μικρομεσαίων. Η κυρία Ριβιέρα Μαντουρέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ κύριε Πίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας μου για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μαζί σας και που είχατε εσείς με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την Επιτροπή μας. Δύο ερωτήσεις να προσθέσω σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Πρώτον, θα ήθελα να μας αξιολογήσετε λίγο πώς λειτουργεί το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Πρόγραμμα πάνω στο οποίο εμείς έχουμε δουλέψει εντατικά. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω για έναν άλλο τομέα της αρμοδιότητάς σας, που είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι μια σημαντική βιομηχανία, σημαντικός κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα, μόνο συντονισμό είχε ως αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα με τη Λισαβόνα θα αυξηθούν οι αρμοδιότητές μας. Έπειτα η οικονομική κρίση επηρεάζει πάρα πολύ τον τομέα. Γι' αυτό και ρωτάω, τι μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιστεύετε ότι μπορεί να ληφθούν ώστε να, δοθούν, να δοθεί νέα όθηση στον τουρισμό και να βοηθήσουμε και με την καινοτομία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ραμστοφ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Είναι μεγάλη χαρά που σας ξαναβλέπουμε εδώ μέσα σήμερα κύριε Πίτροπε. Έχω και μια ερώτηση. Γιατί τις νέες δυνατότητες για, αποθέματα μεθανίου στο permafrost στη Βόρεια Ρωσία. Από ό,τι στοιχεία έχουμε, είναι δυνατόν τα αποθέματα μεθανίου για χρήση να δίνουν διάρκεια 200 με 300 χρόνια από θέματα. Αυτό είναι νέα ανακάλυψη. Και ίσως να επηρεάσει την εξάρτησή μας από τη Ρωσία, να την αυξήσει. Αλλά αυτά τα αποθέματα ως δυνατότητα για το μέλλον έχουν και μία αρνητική πλευρά, δηλαδή με κακή προετοιμασία η χρήση του μεθανίου για παραγωγή ενέργειας να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα μπορούσε ο Επίτροπος να μας πει κάτι παραπάνω για τη νέα αυτή δυνατότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καπόβινσκα. E, Ευχαριστώ. Η συνθήκη της Λισαβόνας κλείνει μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της Ένωσης και μετά για την εφαρμογή των θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Όλοι οι συνάδελφοι σας ευχαρίστησαν κύριε Επίτροπε για τα πέντε χρόνια έργου σας. Εγώ είμαι νεοεκλεγής αβουλευτής και σας συγχαίρω για το ρόλο, σας ευχαριστώ για το λόγο που παίξατε στον ιστορικό αυτό ρόλο της διεύρυνση. Σας ευχαριστούμε, σας ευγνωμονούμε γι' αυτό στην Πολωνή. Η κυρία Χεπέσκα. Ο κύριος. Θα ήθελα να αναφερθώ στη χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη για να στηρίξουμε την καινοτομία. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, να μας πείτε ποιες είναι οι συστάσεις σας προς εμάς αλλά και προς τη Μελλοντική Επιτροπή για να βελτιωθεί αυτός ο μηχανισμός. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος. Συμφωνούμε όλοι καταρχήν ότι η, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων είναι ίδια. Στο κέντρο αυτής της στρατηγικής είναι η ανταγωνιστικότητά μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Όσο πιο βιώσιμη ανάπτυξη έχουμε, τόσο πιο ανταγωνιστικοί θα είμαστε. Γιατί ακριβώς αυτό χρειάζεται σήμερα ο κόσμος. Και νομίζω ότι το θέμα του carbon leakage είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί. Μόνο οι τομείς όπου υπάρχει κίνδυνος έχουν εντοπιστεί και θα υπάρξει εδώ τρόπος να γίνει ένα benchmarking, μια συγκριτική αξιολόγηση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ταξινομηθούν. Αυτή είναι η δική μου, αν θέλετε, κατεύθυνση. Στο τέλος της, αξιολογική, της συγκριτικής αξιολόγησης θα ληφθούν οι αποφάσεις. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και νομίζω ότι συμφωνούμε καταρχήν το είπα εξάλλου και όταν ήταν εκλογές στη Γερμανία. Βέβαια πιο μετριοπαθώς εκφράστηκα εκεί, αλλά σήμερα σας το λέω πολύ απλά. Είναι πολύ δύσκολη η περιβαλλοντολογική πολιτική. Έχουμε ξεκινήσει με δύσκολα βήματα. Σήμερα βεβαίως τα πράγματα έχουν ε, επεκταθεί, υπάρχει κοινή συνείδηση. Όσον αφορά τη συνεργασία που αναφέρατε με χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, αναπτυσσόμενες χώρες, δεν είναι εύκολη η συζήτηση. Και βεβαίως οι δυσκολίες και τα προβλήματα δεν βρίσκονται μόνο στην ευρωπαϊκή πλευρά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δυνατότητες ακόμα Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη πώς εργαζόμαστε και πώς έχουμε οργανωθεί με τις Ηνωμένε Πολιτείες σε ένα επικοδομητικό διάλογο με ευελιξία, με άμεση αντίδραση και πόσο δύσκολα μπορούμε να συνεργαστούμε με την Κίνα που λειτουργεί ακόμα με το Πολιτμπυρό και με ένα κεντρικό σύστημα λήψης αποφάσεων αν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με τους Κινέζους όπως λειτουργούμε με τους Αμερικάνους, θα είχαμε φτάσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα λοιπόν πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία. Στο βασικό ερώτημα που και άλλοι συνάδελφοι έθεσαν, αν το κράτος θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτήν την αλλαγή η απάντησή μου είναι σαφέστατα όχι. Όχι. Και τα κοινωνικά, αν θέλετε, επιχειρήματα δεν αρκούν εδώ. Δηλαδή, για μια επιχείρηση που θα στηρίξουμε, ενώ από υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα και διαρθρωτικές δυσκολίες, στο μέλλον η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Θα είναι ακόμα χειρότερη. Εν πάση περιπτώσει, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης δεν μπορεί να δώσει και δεν προβλέπει ούτε ένα ευρώ για τέτοιου είδους επιδοτήσεις. Ο ρόλος μας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος μας είναι να μην υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοιες δράσεις. Και επαναλαμβάνω, όταν μια τέτοια διαρθρωτική αλλαγή είναι αναπόφευκτη, σκοπός μας και ρόλος μας είναι να τον αναγνωρίσουμε εγκαίρως, να προβλέψουμε και με συνοδευτικά μέτρα να βοηθήσουμε αυτούς που θα πληγούν από αυτήν την διαρθρωτική ε, αλλαγή να βρουν λύσεις. Εγκαίρως λοιπόν, χρόνια πριν συμβεί το κακό αν θέλετε και με επικοδομητικά μέτρα. Σας λέω ότι η άποψή μου είναι να μην παρέμβουμε, είναι πολύ καλύτερο να μην παρέμβουμε εάν είναι κάτι το αμετάκλητο και κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί. Και το λέω αυτό σε όλους τους συναδέλφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα σχήμα στήριξης το οποίο μπορεί να επιτραπεί σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα κρατικής παρέμβασης από μέρους των κρατών μελών εάν, εάν πρόκειται για θέματα που είναι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και δεν έχουν καμία σχέση με ανταγωνισμό προβληματικό μιας επιχείρησης, προβληματική ανταγωνιστικότητα. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο πακέτο μέτρων και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία, η οποία εξάλλου είναι και πολύ απλή. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για πολύ περιορισμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις που οφείλονται, επαναλαμβάνω, αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική κρίση και είναι ε, χρονικά περιορισμένες. Η περίπτωση Opel δεν μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορούμε να σώσουμε καμία επιχείρηση και δεν πρέπει να σώσουμε καμία επιχείρηση η οποία δεν είναι ανταγωνιστική μακροπρόθεσμα. Βράχει πρόθεσμα μπορεί να έχουμε μια μικρή επιτυχία για τις επόμενες εκλογές, αλλά μακροπρόθεσμα η κατάσταση θα είναι χειρότερη. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αν διαγνώσουμε ότι υπάρχει διαρθρωτικό πρόβλημα, πρέπει να μην παρέμβουμε. Κύριε Βάλτσο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι θέμα ούτε των κρατών μελών, ούτε της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Είναι θέμα τραπεζικό. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε κάποια κίνητρα στο τραπεζικό σύστημα έτσι ώστε να υπάρξει ροή και η δανειοδότηση να διευκολυνθεί. Υπήρχε και μια άλλη ερώτηση για το ίδιο θέμα. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέλουμε να προτείνει προγράμματα δανειοδότησης και χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Το κάνει ήδη. Αλλά δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει μικροδιαχείριση εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα κράτη-μέλη έχουν τέτοια προγράμματα και η δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ξέρετε, από ρέων, από μία πρωτοβουλία και χρηματοδοτούνται και από τον δικό μας προπολογισμό. Το μέγεθος των δανείων αυτών βεβαίως μπορεί να επεκταθεί το θέμα των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, όπως ξέρετε. προϋποθέτουν ένα συγκεκριμένο όριο και την ίδια ώρα σήμερα γνωρίζουμε ότι δίνονται κίνητρα σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και πολλούς τομείς όπως την αυτοκινητοβιομηχανία. Πιστεύω ότι στην Ευρώπη, αν κοιτάξουμε όλους αυτούς τους τομείς μαζί, πολύ περισσότερα μπορεί να γίνουν στον τομέα των δανείων. Επίσης έγινε μία ερώτηση για το πρόγραμμα trip για την καινοτομία και το πρόγραμμα Eco Innovation, οικολογική καινοτομία, προγράμματα που θα υποβληθούν στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τα δείτε. Τουρισμός. Την, τετα... την Πέμπτη και την Παρασκευή λαμβάνει χώρα εδώ στις Βρυξέλλες το Φόρουμ με θέμα τον τουρισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρισμό και από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και για πρώτη φορά θα υπάρχουν νομοθετικά εργαλεία γιατί προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από τη χρηματοδότηση κάποιων περιορισμένων προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα αυτού που κάνουμε μέχρι τώρα είναι πολύ θετικά. Αλλά από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνας μπορούμε να κάνουμε πολύ παραπάνω και γι' αυτό και ζητώ ήδη από τώρα από το Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτές τις δυνατότητες. Πρόκειται για ένα από τους πιο σημαντικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, ο τομέας του τουρισμού. είναι ίσως ο μεγαλύτερος τομέας μαζί με την βιομηχανία τροφίμων, ειδών διατροφής, με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Αλλά ακόμα και στον τουρισμό υπάρχουν προβλήματα βιωσιμότητας. Ο ευρωπαϊκός τουρισμός συνδέεται άμεσα με τη μόλυνση, με την καταστροφή της υπαίθρου. Γι' αυτό και πολλοί συνάδελφοι εδώ που ασχολούνται με τον τομέα αυτό ξέρουν πολύ καλά για ποια θέματα ανησυχούμε σήμερα. Υπάρχουν σίγουρα κάποια θέματα που δεν πρόλαβα να τα απαντήσω. Μπορείτε, αν θέλετε, να ζητήσετε και μια γραπτή απάντηση. Σε γενικές γραμμές θέλω να πω όμως ότι με μια γενική πολιτική της νέας κατεύθυνσης στον τομέα της ενέργειας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες και ενδεχομένως το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει μια μαζική μείωση της κατανάλωσης, όποια και να είναι η ενέργεια που χρησιμοποιείται, για περισσότερη αποτελεσματικότητα βεβαίως χρειάζονται μέτρα και επενδύσεις. Το θέμα της προμήθειας είναι ένα θέμα το οποίο δεν λύνει, που δεν είναι λόγο την οικολογική πλευρά της χρήσης ενέργειας. κυρία Κολάνσκα Μπομπίνσκα, δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσατε. Σας ευχαριστώ πάντως. πριν μου δοθεί το όνομά μου σε έναν δρόμο στη Βαρσοβία, θα πρέπει πρώτα να απονείμουμε βραβείο σε εσά, γιατί εσείς είσαστε αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η Πολωνία να γίνει ένα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για τα καλά σας λόγια και για αυτά που είπατε, για το δικό μου ρόλο. Τελειώνοντας, κύριε Πάσκα, βέβαια εδώ χρειάζεται πολιτική πίεση. Εδώ και χρόνια και χρόνια ασχολούμαι με το θέμα αυτό πριν μπω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολύ λίγα έχουν γίνει. Συνεχίζουν να υπάρχουν εμπόδια και αν δεν ξεπεράσουμε τα κοντόφθαλμα εθνικά συμφέροντα και το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δεν προχωρήσουμε σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τότε δεν μπορούμε με τίποτα να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Χρειάζεται λοιπόν πίεση στα εθνικά κοινοβούλια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα το πετύχουμε. Δεν ε, εμποδίζει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας η Επιτροπή. Εμείς έχουμε κάνει πολλές φορές πρόταση. Στο Συμβούλιο κολλάει το θέμα. Και μπορώ απλώς να σας πω, τολμήστε να ξαναφέρετε το θέμα αυτό στο προσκήνιο, γιατί το χρειαζόμαστε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρωστεχνίας. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Ήταν πολλές και πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συνομιλήσουμε. Και ευχαριστώ πολύ. Δεν ήξερα πόσο πολύ χρόνο θα χρειαστούμε. Εγώ πραγματικά μέχρι τελευταίας ημέρας θα υποφεληθώ από αυτήν την συνεργασία μαζί σας. Äh, Κύριε Φερχόγγεν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σίγουρα μας τύχησε μισή ώρα παραπάνω, αλλά νομίζω ήταν απαραίτητο γιατί είχαμε να μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχιστεί η συνεργασία μας. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht weiter. Wir versuchen jetzt ein bisschen. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε την καθυστέρηση που έχουμε. Ο κύριος Ράιμοντ, ο καθηγητής Μπλάχφιτς, ο οποίος θα μας μιλήσει για την οικοκαινοτομία μετά από τη μελέτη που ζητήσαμε και που μας εστάλει μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση στην οθόνη. Έχουμε εδώ φωτοτυπίες της ομιλίας και μπορείτε βεβαίως να την παρακολουθήσετε και να τη διαβάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, χαίρομαι πάρα πολύ και είναι τιμή μου που θα σας μιλήσω σήμερα για το θέμα αυτό. Πριν από μερικούς μήνες κάναμε μια έρευνα. Τα απορίσματα υπάρχουν, μπορείτε να τα διαβάσετε, αλλά θα εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες να τις συζητήσουμε. Τίτλος καινοτομίε. Η Ένωση πώ να μπει σε μια οικονομικά και ενεργητικά αποδοτική οικονομία». Βλέπετε την διάρθρωση και βλέπετε ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο για σπάνι των πόρων. Αυτό είναι σημαντικό για θέματα οικολογικών καινοτομιών. Θα ήθελα όμως να το μελετήσουμε λίγο περισσότερο το θέμα μαζί. Δεύτερο κεφάλαιο είναι το δυναμικό που υπάρχει και ορισμοί. Και τρίτο, πώς να επιταχυνθούν οι οικοκαινοτομίες στην Ένωση. Η σπάνιση λοιπόν των πόρων οι πόροι. Τους τελευταίους μήνες ε, ήρθε λίγο περισσότερο στο κέντρο της δημοσιότητας το θέμα αυτό, γιατί διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη απαιτεί όλο και περισσότερους πόρους. Μπορούν βέβαια να αθρηστούν οι πόροι. Υπάρχει ένα εγκόλπιο της Ένωσης και είναι μια από τις περιοχές του κόσμου η Ένωση όπου τους τελευταίους μήνες και χρόνια απαιτούνται περισσότεροι πόροι. Το ενδιαφέρον στην ιστορία αυτή είναι η αυξανόμενη εξάρτηση από πολλές χώρες προμηθευτές. Όλοι ξέρουμε ότι η Ευρώπη όσον αφορά το αέριο και το πετρέλαιο εξαρτάται πάρα πολύ, 85%. Επίσης, η Ευρώπη και σε θέματα μετάλλων εξαρτάται πάρα πολύ. Σε τέσσερις μεγάλους τομείς εξαρτάται κατά 100% για να καλυφθεί η ζήτηση της βιομηχανίας. Το ίνδιο, το ταντάλιο, το αντιμόνιο, το γάλιο δεν είναι κοινά μέταλλα βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη χαλιβουργία ή για άλλες βιομηχανίες του μέλλοντος. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια διαπιστώνουμε ότι τα αποθέματα είναι μοιρασμένα ισομερώς. Άρα η εξάρτηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα αυξηθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πρόβλεψη για την πιθανότητα της μελλοντική ζήτησης για φυσικούς πόρους. Οι προβλέψεις του ΩΣΑ λένε ότι η ζήτηση για πόρους Πρώτε ύλε, μάλλον θα διπλασιαστεί αν πάρουμε σε βάση το έτος 80. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την Ευρώπη ή από άλλες χώρες του ΩΣΑ. Αυτό έχει σχέση φυσικά κυρίως για τις αναδυόμενες αγορές. Βέβαια, πια έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση όλα, όλα, αν δείτε τις πρώτες ύλες, τις ομάδες πρώτων ύλων, τα βασικά ορυκτά μέταλλα, ενέργεια, βιομάζα, τρόφιμα, παντού, σε όλες αυτές τις πρώτες ύλε, ο σά προβλέπει αύξηση της ζήτησης. Βέβαια, θα διερωτηθεί κανείς ποιες βιομηχανίες θα πληγούν πρώτες. Δεν έχουμε know-how. Χρειαζόμαστε ένα ραντάρ κινδύνου στην Ένεση για να μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες βιομηχανίες ακριβώς στα επόμενα χρόνια θα χρειαστούν ποιες πρώτες ύλες. Αυτό το know-how δεν υπάρχει. Πάντως το ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν όλες οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας απαιτούν πρώτες ύλες, ιδιαίτερα τα κρίσιμα μέταλλα. Παραδείγματος χάρη, τα κινητά, τις επίπεδες οθόνες που έχουμε στους υπολογιστές, η συζήτηση που γίνεται εδώ με τα μικρόφωνα και λοιπά, Αυτό που συζητήσετε πριν για τα αυτοκίνητα, όλα αυτά απαιτούν αυτά τα μέταλλα. Έπειτα το μέλλον της βιομηχανίας είναι πράσινο, ακούσαμε. Σωστό. Αλλά και οι πράσινες βιομηχανίες και τεχνολογίες απαιτούν αυτά τα μέταλλα. Τα χρειάζονται για τον τριμερή καταλήτη, για την αιωλική ενέργεια, για την σύζευξη πηγών ενέργειας, για το αυτοκίνητο που θα λειτουργεί με υδρογόνο ή το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όλοι αυτοί, όλες αυτές οι τεχνολογίες απαιτούν αυτά τα μέταλλα. Ένα επιχείρημα λέει ότι η αύξηση στην αποδοτική παραγωγή αυτών των πρώτων υλών είναι ένας τρόπος να βγει να προχωρήσει η Ένωση. Βέβαια, αν συγκριθούμε για την παραγωγικότητα των πρώτων πώς αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την παραγωγικότητα της ενέργειας ή της εργασίας. Ε, είμαστε πιο εργατικοί, αυξήθηκε η αποδοτικότητα της εργασίας. Η αποδοτικότητα όμως των, στις πρώτες ύλε υστερεί. Ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε τους, τα παλιά κράτη-μέλη, τους 15, με τις νέες χώρες μέλη Ένωσης βλέπουμε νέους αριθμούς Βλέπετε τα πιο πρόσφατα νούμερα. Διεπιστώνεται ότι η παραγωγικότητα της ενέργειας και της εργασίας στις νέες χώρες μέλη είναι, εξηγήστε πολύ θετικά, η παραγωγικότητα στην αφορά τις πρώτες ύλες υστερεί, για διάφορους λόγους. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το δυναμικό είναι πιο μεγάλο, προκειμένου η αποδοτικότητα της πρώτης ύλης βραχυπρόθεσμα και στις χώρες αυτές να αυξηθεί. Η απέτηση της Ένωσης η Ευρώπη να γίνει η πιο αποδοτική όσον αφορά σε πρώτες ύλες οικονομία του κόσμου δεν είχε ακόμα επιτευχθεί. Η σπάνιες λοιπόν των πρώτων υλών είναι ένα ερώτημα κλειδί. Όχι για το μακρινό μέλλον, για το άμεσο μέλλον. Για πολλές βιομηχανίες. διατραζώντας την χρηματοπιστωτική κρίση έχουμε έναν ορισμό της, των οικοκαινοτομιών που αναφέρει ότι οι οικοκαινοτομίες είναι σημαντικές για ε, μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, αλλά και όσον αφορά την αποδοτική χρήση των πρώτων υλών. Και πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο μικρό επίπεδο, το επίπεδο της επιχείρησης, το επίπεδο διαφόρων αλυσίδων, όλης ροής των πρώτων υλών πάμε σχετικά τι συμβαίνει με, το χάλιβα, με, τον, ε, με τον χαλκό διεθνώ και με τη γενική οικονομία της Ένωσης. Αν δούμε ποιος έδρασε τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτική χρήση των πρώτων λόγων, είναι πολλές επιχειρήσεις παραγωγικές. Δηλαδή, προσπάθησε ο καθένας μέσα στον χώρο του το κόστος των υλικών να μειωθεί και υπήρχε σχετική επιτυχία. Αυτό που ακόμα δεν έχει αυξηθεί είναι το δυναμικό του μέλλοντος. Αυτό υπάρχει και downstream και upstream όσον αφορά την παραγωγή πρώτων υλών, τη χρήση των πόρων αυτών. Για ποιους τομείς μιλάμε που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση μεταξύ των ε, οικονομοβόρων βιομηχανιών και των πρώτων ελληνών βόρων βιομηχανιών. Είναι οι κατασκευές, η κινητικότητα, τρόφιμα και ποτά. Επόμενο slide. Συγκεκριμένα παραδείγματα όπου μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι οικοκαινοτομίες είναι δυνατόν να υλοποιηθούν συγκεκριμένα. Θα δω μόνο στα κτίρια. Θα έχει ακούσει το Zero Emission, Low Carbon, διάφορες προσπάθειες στα σπίτια μας. Να καταλήξουμε σε χρήση ενέργειας μηδέν είναι δυνατόν ή να συνδεθούμε με διάφορα δίκτυα. Αυτό θέλουμε να το επεκτείνουμε με οικοκαινοτομίες. που λαμβάνει υπόψη την, ε, ε, την παράμετρο χρήσης πρώτων υλών για την ενέργεια. Να έχουμε ένα functional integrated envelope, δηλαδή να υπάρχει ένα είδος συνολικού φακέλου όσον αφορά την κάλυψη του κτηρίου. Ένα συγκεκριμένος τύπος οικίματος. Ωστόσο, Πάντα στον τομέα αυτό δεν μπορεί τα πράγματα να γίνουν από μόνο τους. Χρειάζονται πολλοί φορείς. Αλλά υπάρχουν και πολλά εμπόδια. Εδώ συγκεκριμένα είναι το θέμα εκμισθωτή-μισθωτή, τα, ο χρόνος payback, δηλαδή ποιος ε, ιδιοκτήτης θα υπολογίσει πόσο χρόνο για 10 χρόνια και επιπλέον. Πώς θα γίνει δηλαδή η αποπληρωμή ορισμένων επενδύσεων η απόσβεση μάλλον ορισμένων επενδύσεων. Εδώ, είδη διατροφής, αποθήκες, διάφορες ε, οικοκαινοτομίες που μπορούν να γίνουν σε αποθήκες ειδών διατροφής. Στο επόμενο slide βλέπετε πάρα πολλά εμπόδια και επίσης και τους θετικούς φορείς οι οποίοι θα διακινήσουν την νέα αυτή διάσταση. Ας δούμε την παγκόσμια αγορά. Μια νέα μελέτη της Roland Berger σε μια μελέτη της Σιρόνα Μπέργκερ μας λέει ότι η παγκόσμια αγορά είναι πράσινη. Ποσοτικά αυτό σημαίνει ότι σε όγκο για τις οικοκαινοτομίες στα επόμενα 10 χρόνια θα διπλασιαστεί. Δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης σε αυτό το τομέα είναι πιο, πολύ, πιο μεγάλος από ό,τι σε άλλους τομείς της βιομηχανίας. Η αγορά για πρώτες ύλες και αποδοτική χρήση τους κατά πάσα πιθανότητα θα τριπλασιαστεί μέχρι το 2020 και συνολικά ο όγκος αγοράς για οικοκαινοτομίες ανάγεται σε 3-3 ευρώ. Το θέμα είναι πώς οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, όχι μόνο στην Ευρώπη, να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα αυτά επεξεργαζόμενοι και μια διεθνή στρατηγική. Υπάρχουν και εμπόδια. Και εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος του πολιτικού. Όχι μόνο για το θέμα της ρύθμισης, αλλά να υπάρξει μια πολιτική που να έχει στόχο την ικανότητα της αγοράς να αυξήσει την πληροφόρηση των πολιτών και να αξιοποιήσει το δυναμικό οίκο καινοτομιών. Επόμενο slide. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που προσπαθούν να προωθήσουν οικοκαινοτομίες. Παραδείγματο χάρη, η δυνατότητα του eco-design, η οδηγία για το eco-design, Το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, ε, το πρόγραμμα δράσης για την ε, τεχνολογία περιβάλλοντος, ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, όλα αυτά σε επιμέρους τομείς προσπαθούν να αξιοποιήσουν το δυναμικό οικοκαινοτομιών. Βέβαια, ακόμα υπάρχουν ορισμένα στρατηγικά κενά. Πάμε σε μια εφεύρεση. Πώς περνάει από τον εγκέφαλο του ερευνητή μέσω του γκαράζ στην αγορά. Δηλαδή κάθε καλή ιδέα δεν καταφέρει να φτάσει πάντα μέχρι την αγορά. Έπειτα έχουμε ένα δεύτερο χάσμα, εκεί που ένα πρωτότυπο, ένα πρότυπο λειτουργεί, μεν, αλλά για να φτάσει στη μαζική παραγωγή χρειάζεται πάρα πάρα πολύς χρόνος. Και εδώ έχουμε δύο στρατηγικά κενά, για τα οποία η εθνική πολιτική και η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να είναι πιο παρούσα, έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό. Αν δείτε τα διάφορα προγράμματα σχετικά με τα κενά αυτά και τις ευκαιρίες τα βλέπετε στο διάγραμμα. Και άλλα παραδείγματα εδώ, περνάω στα γρήγορα, περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Τι, τι είναι το πρακτέον. Ένα από τα πορίσματα είναι να υπάρχουν κίνητρα που να στηρίζονται στην αγορά, εργαλεία που να στηρίζονται στην αγορά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στον τομέα αυτό επιπλέον των διαφόρων προσπαθειών στην ενέργεια. Παραδείγματο χάρη το εμπόριο εξατμίσεων, εκπομπών δηλαδή, τη σχετική οδηγία. Θα μπορούσε η Ευρώπη να κάνει να φορολογήσει παραδείγματο χάρη υλικά που χρησιμοποιούνται για κατασκευέ. Οι μισέ χώρε το κάνουν. Έτσι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα στη χρήση αυτών των πρώτων υλών στις κατασκευές. Μετά έχουμε την περιφερειακή πολιτική. Περίπου το 80% των δαπανών πάνε για τη γεωργία και τα περιφερειακά προγράμματα. Η δράση και η στα κονδύλια αυτά μπορεί να αυξηθεί και κάνουμε και μερικές προτάσεις. Και αυτό έχει σχέση με καινοτομίες που μπορεί να ε, εισαχθούν στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Έχει το πρόγραμμα δράσης για την βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη κατανάλωση και άλλα παρόμοια. Επόμενη διαφάνεια. Η βιομηχανία προς το συμφέρον της θα πρέπει να φροντίσει να μειωθεί το κόστος πρώτων υλών. Η βιομηχανία βλέπει τους κινδύνους μια τέτοια, που συνδέεται με μια τέτοια ριζοσπαστική πολιτική καινοτομιών. Εμείς δίνουμε τις διάφορες δυνατότητες. Στην αρχή έχουμε μια στρατηγική που στοχεύει στη μείωση του κόστους των πρώτων υλών. Μετά έχουμε άλλες στρατηγικές με τις οποίες η βιομηχανία τους ζητάει από τους πελάτες αποδοτική χρήση των πρώτων υλών και εξοικονόμηση. Μετά έχουμε στις, ε, στις υπηρεσίες και στις καινοτομίες. Έπειτα οι επιχειρήσεις πώς μπορούν να χρησιμοποιούν νέα πακέτα υπηρεσιών ή να τα πουλάνε. Βέβαια υπάρχει και μια ανάγκη για νέες καινοτομίες, νέες πρωτοβουλίες. Αναφέρονται και αυτά στη μελέτη. Η χρηματοδότηση οικοκαινοτομιών στην Ευρώπη μέχρι στιγμής υστερεί. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρχει ένα ταμείο ευρωπαϊκό ειδικά για την πρόθεση των οίκο-καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Από όπου μια επιχείρηση να μπορεί να πάρει κεφαλαία κινδύνου. Υπάρχει πρότυπο γι' αυτό. Στην Αγγλία υπάρχει αυτό για τον άνθρακα, Carbon Trust Fund το λένε εκεί, το οποίο επιδείχθη ιδιαίτερα επιτυχές για τον άνθρακα. Ας διδαχτούμε από αυτό το καλό παράδειγμα να κάνουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, ένα τέτοιο ταμείο. Δεύτερο σημαντικό τομέα είναι η κοινοτομία των υλικών. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια τεχνολογική πλατφόρμα για τις βιομηχανίες κατασκευές, Φερρυπίν, όπου έχουμε τα υλικά, στα επιστημονικά στοιχεία, έχουν πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες κατασκευών και τα αυτοκίνητα, γιατί ένα αυτοκίνητο ζυγίζει πάνω από ένα τόνο πολλές φορές. Αν λοιπόν μειωθεί το υλικό με την ηλεκτροκινητικότητα ή άλλες μορφές ε, του οχήματος που έχει εκπομπές μηδέν, αυτό θα ήταν ωφέλιμο. Και το τρίτο, ένα πρόγραμμα καινοτομία όσον αφορά τα κτίρια. Ξέρετε ότι όλες οι χώρες μέλη του ζητήθηκε να εφαρμόσουν την οδηγία αποδοτικής χρήσης της ενέργειας για τα κτίρια. Οδηγία. Καλό θα είναι αν θέλουμε να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία και να διδαχθούμε από τις πρωτοπόρες χώρες, σιγά σιγά να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βαθμία για την ανακαίνιση των κτηρίων ενεργειακά ενώ, με στόχο να μειωθούν και εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και να αυξηθεί η αποδοτική χρήση των πρώτων υλών. Και με αυτό τελείωσα. Η τελευταία μου διαφάνεια σας λέει ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος, ο κύριος Τόμας, έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να μπούμε μέσα σε αυτή τη μελέτη και να εξετάσουμε κάποιες άλλες πτυχές και ο κύριος Φερχόγγι νομίζω θα συμφωνήσει ότι το θέμα του περιβάλλοντος, το θέμα των πόρων θα πρέπει να δώσει νέες ε, ευκαιρίες και δυνατότητες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Δηλαδή να μην βλέπουμε αυτές τις επενδύσεις σαν επιπλέον δαπάνες, αλλά σαν επιπλέον ευκαιρίες. Τρία σημεία θα ήθελα να θίξω. Πρώτον, μιλήσατε για αυτά τα gaps, τα χάσματα όσον αφορά την πολιτική καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρατε δύο χάσματα, δύο κενά. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί υπάρχουν ακόμα εμπόδια σε αυτή την πολιτική κοινωνία. Δεύτερον που θα ήθελα να μάθω. Πού υπάρχει η ισορροπία μεταξύ ρύθμισης, δηλαδή αυστηρή νομοθεσία για απόβλητα, για λύματα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Έχουμε αποδείξεις για την σχέση μεταξύ αυστηρής νομοθεσίας και κινήτρων, γιατί χρειαζόμαστε αυστηρή νομοθεσία, παραδείγματο χάρη για τα νέα κτίρια, έτσι ώστε να στραφεί η αγορά προς την καινοτομία. Αυτά, αυτά τα δύο ήθελα να ρωτήσω και φαίνω το λόγο του επόμενου. Ευχαριστώ, κύριος Μπίτελγκόφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Τόμας και να κάνω κι εγώ δύο ερωτήσεις προς τον καθηγητή. Προετοιμάσατε μία έκθεση για μας Και το θέμα της αποτελεσματικότητας των πρώτων υλών, των φυσικών πόρων και της ενέργειας, βλέπουμε ότι αν κάνουμε μία ε, σύγκριση της καλύτερης και της χειρότερης απόδοσης, πάμε από το 1 στο 17. Ερωτώ λοιπόν, τι τρόπο μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βοηθήσει τις χώρες που είναι οι πιο απομακρυσμένες από την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και αυτή η νέα καινοτομία και στρατηγική καινοτομία πώς μπορεί να συμπεριλάβει και όλα τα κράτη τα οποία είναι ίσως και τα πιο καθυστερημένα και να μην απευθύνεται μόνο στα πιο αναπτυγμένα κράτη. Δεύτερη ερώτηση πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λάβουμε υπόψη μας πως άλλοι οικονομικοί χώροι και άλλες χώρες θεσπίζουν και υλοποιούν στρατηγικές στον τομέα της καινοτομίας, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποια είναι τα παραδείγματα τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν στους άλλους οικονομικούς χώρους. Υπάρχουν σε κάποια σημεία και πιο αποτελεσματικές στρατηγικές από τη δική μας. Ευχαριστώ κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ. Φαίνεται σαν είναι μια πράσινη συζήτηση, αλλά τι να προσθέσω μετά από αυτά που είπε ο συνάδελφο. Ήταν οι ερωτήσει που ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Όπω επίση και για το θέμα τη εξοικονόμηση ενέργεια. Οπότε τίποτα δεν έχω να προσθέσω. Ο κύριο Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ακριβώ αυτό που είπε και ο προηγούμενο συνάδελφο όταν μίλησε ε, στον Επίτροπο, τον κύριο Φερχόγγεν. Μίλησε για μια κατευθυντήρια γραμμή, για μια ιστορία. Και θα πετύχουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιομηχανία παρά μόνο εάν ενσωματώσουμε καινοτομία και καινοτόμες δράσεις. Τώρα, στην παρουσίασή σας και στην παρουσίαση της κάθε πολιτικής σε αυτό το τομέα υπάρχουν κάποιες ιδεολογικές κατευθύνσεις και διαφορές. Παράδειγμα, η αυτοκινητοβιομηχανία. Τι μπορούμε να εντοπίσουμε σαν οικολογικές καινοτομίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και το ερώτημα είναι αν μια καινοτομία είναι οικολογική ή όχι. Ξέρετε ότι σήμερα δόθηκε το βραβείο Νόμπελ και δόθηκε για τις οπτικές ίνες. Κάτι δηλαδή που ανακαλύφθηκε στη δεκαετία του 60. Τα καλώδια οπτικές ίνες δεν είναι καινούριο. Βλέπετε όμως ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή αυτή η καινοτομία είναι και οικονομικά, οικολογικά συγγνώμη, βιώσιμη, μειώνονται οι εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα, είναι και οικολογική καινοτομία. Εσωτερικά λοιπόν των διαφόρων αξιολογήσεων και στο εσωτερικό της Επιτροπής πολύ συγκεκριμένα υπάρχουν οικολογικές καινοτομίες που αγνοούνται για ιδεολογικούς λόγους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει μόνο στο χαρτί τι είναι η κάθε καινοτομία και πιστεύω ότι εδώ μια τεχνική διαδικασία που έχουμε, που είναι η επιτροπολογία, θα πρέπει να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτές τις ιδεολογικές διαφορές. Και οι οικολογικές καινοτομίες θα πρέπει να προχωρούν απρόσκοπτα και να υλοποιούνται. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόμσον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι μέλη της Επιτροπής μας. Στο προηγούμενο κοινοβούλιο εγκρίναμε μια οδηγία για μείωση 20%. όσον αφορά τη βιώσιμη ενέργεια και μία εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 20%. Αυτή ήταν δεσμευτική η στόχη. Αν δεν περιορίσουμε την κατανάλωση της ενέργειας, θα πράττουμε συσήφιο έργο. Θα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο ενέργεια. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν σε εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτική χρήση της ενέργειας. Γι' αυτό οι οικοκαινοτομίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Μερικά παράδειγμα από τη Δανία. Προσπαθούμε ο κόσμος στον χώρο εργασίας του να, να υιοθετεί μεθόδους καινοτομία όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτική χρήση της. Κυρίως όμως το πρόβλημα θεωρώ είναι ότι όταν δούμε την οδηγία αυτή για τις ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση του διοξείδιου του άνθρακα, χρειαζόμαστε δύο δεσμευτικούς στόχους. Το είπε και η Άγγελα Μέρκετ. Χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους για τη βιομηχανία γιατί η βιομηχανία θα επενδύσει μόνο μα έχει δεσμευτικούς στόχους. Εδώ μιλάμε για αποδοτική χρήση της ενέργειας και εξοικονόμηση. Ε, λοιπόν, γι' αυτό δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι. Πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους. Πρόεδρος. Άλλος. Ζαντό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση στον καθηγητή. Μας έδωσε ένα πολύ ε, σαφές πλαίσιο, Υπάρχει, δεν υπάρχουν ανακολουθίες. Το ερώτημα είναι το εξή. Τι λείπει από το πακέτο ενέργεια περιβάλλον έτσι ώστε είτε για τα κτίρια είτε για το eco-design να μην πετυχαίνουμε συγκλίνοντες στόχους. Απλή ερώτηση. Επαναλαμβάνω. Με στόχο μείωση κατά 20% της κατανάλωσης του 2020 που να μην είναι δεσμευτικό είναι δυνατόν να πετύχουμε ε, μέτρα τα οποία μεταξύ τους να συμφωνούν όσον αφορά τις οικοκαινοτομίες. Γκίρεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά της ε, οικοκαινοτομίας υπάρχουν και άλλες λύσεις συναφείς σχετικά με την μείωση μάλλον σχετικά με την χρήση της ενέργειας και τη σχετική μείωση. Το θέμα αυτό ακόμα δεν έχει μελετηθεί σε βάθος. Κάτι σημαντικό όμως είπε ο κύριος καθηγητής ο θερμικός εξυγχρονισμός είναι η κύρια έρευνα που σχετίζεται με τις οικοκαινοτομίες, το κύριο μέτωπο. Εγώ γι' αυτό θα κάνω μια γενική παρατήρηση. Ο στόχος 20-20-20 είναι σωστός και φιλόδοξος και θα επιτευχθεί μέσω του πακέτου ενέργεια-κλίμα. Κάθε χώρα θα πρέπει να εφαρμόζει με τον ίδιο τρόπο, αλλά οι συνθήκες από χώρα σε χώρα διαφέρουν. Αυτές εδώ οι καινοτομίε, κατά κάποιο τρόπο, ανάλογα με τις προτεραιότητε, θα πρέπει να εφαρμόζονται. Οι προτεραιότητες όμως δεν έχουμε. Πάμε χάρη στη χώρα μου την Πολωνία, που χρησιμοποιεί τον άνθρακα ω πηγή ενέργεια κυρίω η εφαρμογή τη λύση που να έχει σχέση με τον άνθρακα μπορεί να είναι χρήσιμη. Ο εξυγχρονισμό των κτηρίων θα μα οδηγούσε σε περισσότερη εξοικονόμηση όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι προβλέπει το φιλόδοξο πρόγραμμα 2020-2020. Κανείς άλλος δεν ζητάει το λόγο. Το λόγο στον κύριο καθηγητή για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις πραγματικά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες και ελπίζω καταρχήν να απαντήσω στο ερώτημα πώς ξεχωρίζει κανείς τις οικολογικές καινοτομίες. Τι είναι οικολογικές καινοτομίες? Οι οικολογικές καινοτομίες πρέπει να ειδωθούν υπό ένα παγκόσμιο πρίσμα, αν θέλετε, και αν συνεχιστούν οι προσπάθειες στην Ευρώπη για την χρήση των συσκευών ή των αυτοκινήτων, Ακούσαμε σοβαρή κριτική τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα βιοκάψιμα. Ότι ναι, είναι καλή η πρόθεση, αλλά υπάρχουν χώρες, όπως αναπτυσσόμενες χώρες, που παράγουν τόσο εντατικά αυτά τα βιοκάψιμα, έτσι ώστε τα τελικά τα μειονεκτήματα είναι περισσότερα από τα πλεονεκτήματα. Γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε λίγο πιο μακρυπρόθεσμα και σφαιρικά τέτοιες οικολογικές καινοτομίες και δεν είναι εύκολο να τα αξιολογήσουμε σφαιρικά. Υπάρχουν σήμερα τρόποι όπως το portfolio management, την οικολογική αξιολόγηση, Υπάρχουν τρόποι αξιολόγησης αυτών των οικολογικών καινοτομιών. Μια μικρή επιχείρηση η οποία είναι στραμμένη προς την καινοτομία έχει δυσκολία να κάνει αυτή τη σφαιρική αξιολόγηση και θα πρέπει να στηριχθεί σε εξωτερικούς φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς για να κάνει αυτή την οικολογική αξιολόγηση. Στόχοι πόσο δεσμευτική πρέπει να είναι, πόσο αυστηρή πρέπει να είναι η στόχη που θέτουμε. Πιστεύω ότι όσον αφορά την οικολογική καινοτομία, θα πρέπει να θέσουμε ένα μακροπρόθεσμο στόχο και προσανατολισμό. Παραδείγματο χάρη για την αλλαγή του κλίματος έχουμε θέσει τέτοιους στόχους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μακροπρόθεσμους στόχους έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος, αλλά και οι επιπτώσεις επί των επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από αυτές οι οικολογικές καινοτομίες πραγματικά θα πρέπει να ειδωθούν με μια προοπτική 20-30 ετών. Ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί με υδρογόνο παραδείγματο χάρη, που είναι η νέα λύση που συζητείτε. 20 χρόνια τουλάχιστον μέχρι να το δούμε στους δρόμους της Ευρώπης. Τίθενται λοιπόν στόχοι ύψης της προτεραιότητας και μιλάμε για το 2020, 50 και κατόπιν γίνεται μια ταξινόμηση, μια ε, ιεράρχηση όσον αφορά τη δεσμευτικότητα αυτών των στόχων. Η αυστηρότητά τους, αν θέλετε, και η δεσμευτικότητα αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός. Ρωτήσατε επίσης τι ρύθμιση είχε επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Οι οδηγίες όντως οδήγησαν σε πολλές καινοτομίες. Η αλήθεια είναι όμως ότι μια τέτοια ρυθμιστική πολιτική αυξάνει το, τη γραφειοκρατία, άρα έχει και αρνητικά σημεία όσον αφορά την καινοτομία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με αυτές τις καινοτομίες. Η πρόσβαση στην πληροφορία για τα υλικά, παραδείγματος Σήμερα δεν υπάρχει παρά μόνο ένας οργανισμός, το Eurogeo Survey, που δίνει πληροφορίες όσον αφορά την ζήτηση των πρώτων υλών στην Ευρώπη. Μας λείπει λοιπόν ένα είδος τράπεζας δεδομένων που δίνει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που το επιθυμούν. Δεύτερον, πληροφορίες επί των ίδιων των προϊόντων. Πολύ σημαντική πρόοδος έγινε όσον αφορά το carbon footprints και αυτό που λείπει είναι ένα ευρωπαϊκό σήμα για τα προϊόντα και τις πρώτες σύλλες σε σχέση με τον αντίκτυπο του άνθρακα. Δεν πρέπει βέβαια να επικεντρωθούμε μόνο στο διοξίδιο του άνθρακου, αλλά γενικότερα την χρήση κάποιων πηγών ενέργειας και τα αποτελέσματα επί του περιβάλλοντος, τον αντίκτυπο επί του περιβάλλοντος. Ζητήσατε επίσης πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Από το 1 στο 17 είπατε. Η πιο αποτελεσματική χώρα χρησιμοποιεί το 1 δέκατο προϊόντων και αυτά πάντα σε σχέση με το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Έχετε δίκιο λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τι μπορούν να κάνουν χώρες με χαμηλή αποτελεσματικότητα. Οι νέε χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία. Δεν ξέρω. Και βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και μετά την οικονομική κρίση όταν οι επενδύσεις αρχίζουν να γίνονται πιο στοχευμένα σε τομείς και σε συγκεκριμένες καινοτομίε. Τα δημόσια κτίρια, παραδείγματο χάρη, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα παράδειγμα για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Αλλά και τα ιδιωτικά κτίρια, οι επενδύσεις, τις μεταφορές. Όλοι αυτοί οι τομείς προσφέρουν δυνατότητες για καθοδήγηση των επενδύσεων σε τομείς που προσφέρουν δυνατότητες οικολογικής καινοτομίας. Carbon leakage. Αυτό είναι ένα θέμα που σαφώς και παρατηρείται εντονότατα στα νέα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εγκαταστάθηκαν βαριές βιομηχανίες. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να προτείνουμε πακέτα μέτρων στη χαλιβουργία, στην τσιμεντοβιομηχανία, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδόσεις αυτών των βιομηχανικών τομέων. Και σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης, με ρωτήσατε τι παραδείγματα υπάρχουν στην Ευρώπη, αλλά και εκτός της Ευρώπης. Υπάρχουν παραδείγματα. Η Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη. Είναι η πιο αποτελεσματική χώρα όσον αφορά την εξοικονόμηση και χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων. Η Ιαπωνία εδώ και πολλά χρόνια ενσωματώνει καινοτομίες με πολλές οικολογικές επιπτώσεις στην πολιτική της και από την Ιαπωνία πολλά μπορεί να μάθει η Ευρώπη. Τα αποτελέσματα είναι καλά. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στην Κίνα. Η μεγαλύτερη ζήτηση για άνθρακα, για πετρέλαιο, προέρχεται από την Κίνα. Την ίδια ώρα όμως, η πολιτική της Κίνας για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι θεματική. Επίσης, το ίδιο μπορούμε να πούμε και για άλλους τομείς, όπως οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια η Κίνα μπορεί να δημιουργηθούν κέντρα στην περιοχή της Σανγκάη, παραδείγματο χάρη, με μηδανικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και μπορεί να γίνουν πρότυπα και μοντέλα για άλλες ασιατικές περιοχές και πόλεις. Και εμείς οι καλοί Ευρωπαίοι τι κάνουμε σε σχέση με αυτές τις χώρες, τις αναπτυσσόμενες χώρες ή την Ιαπωνία. Όντως η Ευρώπη θα πρέπει να προσπαθήσει να μην χάσει το τρένο. Ξέχασα κάτι. Ναι, κύριε Τόμσον, μιλάτε για την Δανία. Ναι, όντως υπάρχουν κάποια στοιχεία για τη Δανία, για όλες τις σκανδιναβικές χώρες, με πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα, σίγουρα, όσον αφορά τις οικολογικές καινοτομίε. Μιλήσατε και για τα κενά, κύριε Τόμψον. Ποιες είναι οι κύριες αδυναμίες Ναι, έλλειψη πολλές φορές τόλμης από μέρους των επιχειρηματιών και από μέρους των επενδυτών. Ε, όντως αυτό πλήττει και την οικολογική καινοτομία, όχι μόνο την καινοτομία. Είναι φοβισμένοι οι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν πολλές καλές ιδέες, τολμηρές ιδέες, οι οποίες δεν προχωρούν. Η Ιαπωνία είναι πολύ καλή σε αυτό το τομέα ότι από το ξεκίνημα μια καλή ιδέα μέχρι τη διάθεση αγοράς ενό προϊόντο περνάει πολύ λιγότερο χρόνο. Εμεί, λοιπόν θα πρέπει εδώ να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Και γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος βελτίωσης, πολλές προτάσεις που συζητούνται και οι οποίες θα πρέπει να μας οδηγήσουν προ αυτή την κατάσταση. Έχουμε δυνατότητε, αλλά θα πρέπει αυτό το δυναμικό να οδηγήσει σε συγκεκριμένες και απτές καινοτομίες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπλάισβιτ, για τις πληροφορίες σας, τα στοιχεία που μας δώσατε, αλλά και για τη δυνατότητα που μας δώσατε να κάνουμε ερωτήσεις και να εμβαθύνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι τελειώσαμε και με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Kollege Thomas. Vielleicht noch für die neuen Kollegen wäre es noch gut zu wissen. Για τους νέους συναδέλφους, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε πού υπάρχουν αυτά τα έγγραφα. Πού μπορεί κανείς να βρει αυτή την έρευνα, αυτή τη μελέτη. Wir werden eine Rundinformation machen. An alle. Einverstanden? Ναι, ναι, θα δώσουμε τις πληροφορίες με mail. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή αποδομή εντό της ευρωπαϊκή Κοινότητας. Δεν είναι παρόν ο εισηγητή. Ο κύριος Όλο η κυρία Όλ θα πάρει το λόγο. Κύριε Χάουλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την ειλικρινή συγνώμη της κυρίας Βαλεάν που δεν είναι εδώ σήμερα. Δεν μπόρεσε να έρθει στις Βρυξέλλες. Αναρωτιέμαι λοιπόν Μήπως θα βοηθούσε αν δίνατε το λόγο πρώτα στην Κομισιόν για να μας πούνε τις απόψεις τους και μετά να κάνουμε εμεί ό,τι ερωτήσεις και σχόλια έχουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση δηλαδή. Γίνεται αυτό. Ναι, ο Πρόεδρος. Δεν ξέραμε ότι δεν θα ερχόταν εδώ η συγγήτρια, οπότε εντάξει, αν δεν έχει αντίρρηση η Επιτροπή, ξεκινήσει εκείνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση ενέργεια από την Κομισιόν. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει την πρόταση αυτή όσον αφορά κανονισμό για την διόρθρωση όσον αφορά τις υποδομές τις ενεργειακές. Γιατί πιστεύουμε ότι σε 10-15 χρόνια θα έχουμε μια αποφασιστική στιγμή για κάθε είδους απόφαση που θα πάρουμε για τις ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη. Οι ενεργειακές υποδομές, είτε πρόκειται για το πετρέλαιο, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε πρόκειται για την προήθεια, είτε για την παραγωγή, είτε για την μεταφορά ενέργειας, πρόκειται για υποδομές οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν μεγάλο κύκλο ζωής και ό,τι επενδύσεις γίνουν σήμερα θα εξακολουθούν ε, να αποφέρουν καρπούς και μετά από 30-40 χρόνια. Είναι λοιπόν αποφασιστική σημασία να ξέρουμε η Ευρώπη θα μπορέσει να έχει ένα ενεργειακό μείγμα που να ελαχιστοποιεί τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και βασιζόμενοι στο γεγονός ότι το, η ατμόσφαιρα επενδύσεων δεν είναι και η καλύτερη δυνατόν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι κάθε δύο χρόνια για παράδειγμα βάσει συγκεντρωμένων στοιχείων από τα κράτη-μέλη να μπορούμε να αξιολογούμε τις επενδύσεις που γίνονται και την κατάσταση γενικότερα για να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις υποδομές της ενεργειακές στην Ευρώπη που προβλέπεται κάποιο τέτοιο πρόβλημα είτε πρόκειται για τον ηλεκτρισμό είτε για το φυσικό αέριο είτε για κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να βασιστεί στον κανονισμό του 96 που αυτός με τη σειρά του βασίζεται σε άλλες αποφάσεις της δεκαετίας του 70 να εξυγχρονίσουμε λοιπόν αυτή τη ρύθμιση που έχουμε στη διάθεσή μας. Τι έχουμε υποβάλει μέχρι τώρα. Προτείνουμε κάθε δύο χρόνια, όπως σας είπα, τα κράτη-μέλη να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδομένα όσον αφορά τις δυνατότητες που προβλέπουν να έχουν, τι υποδομές σχεδιάζουν στον τομέα του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επίσης και να μας μιλήσουν για την αποθήκευση και την μεταφορά διοξιδίου του άνθρακα. Δεν θέλουμε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Εμείς δεν αποτελούμε γραφείο σχεδιασμού. Οι υποδομές έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που διαχειρίζεται ο κλάδος. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι δεδομένων των στόχων που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα θέλαμε να γνωρίζουμε κι εμείς αν όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια, τι δυνατότητες υπάρχουν, τι θα προσθεθεί, ποιες είναι οι προθέσεις που έχουν διάφορες χώρες στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουν καθορίσει. Μερικές φορές χρειάζεται περισσότερος χρόνος για κάποιους λόγους. Όλα αυτά θέλουμε να τα αναλύσουμε και να τα αναλύουμε κάθε δύο χρόνια. Μερικές φορές πρόκειται για καθαρά οικονομικά δεδομένα, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι περιορισμένη η πρόσβαση σε επιστώσεις ή να υπάρχουν εμπόδια στον σχεδιασμό σε ορισμένες χώρες μέλη. Ή ακόμα μπορεί να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ε, πράγματα τα οποία συνδέονται με την κατάσταση στην τοπική αγορά. Η πρόταση λοιπόν που εξετάζει η συγγήτριά σας, βλέπουμε ότι μιλάει για το τι ήδη υπάρχει και τι, θα, τι προβλέπετε. Και μας ρωτάει η συγγήτρια γιατί κάθε δύο χρόνια. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται αυτό, μια που πρόκειται και για συναπόφαση από πλευρά του Κοινοβουλίου. Οπότε κάθε δύο χρόνια πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιολογείται η κατάσταση για να γίνεται καλύτερη διαχείριση του δικτύου και των υποδομών. Δεν θα υπάρχει μεγάλο διοικητικό άχθος. Θέλουμε να υπάρχει μια συνοχή με τα μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Θέλουμε επίσης κάθε δύο χρόνια να μας λένε τα κράτη-μέλη τι ισχύει και όσον αφορά άλλες δυνατότητες ενεργειακές που έχουν Αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύει αυτά τα δεδομένα. Είναι κάτι που εξάλλου αδιάκοπα ζητάει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επίσης θέλουμε και προβλέψεις στον τομέα της κατανάλωσης για να μπορούμε να συγκρίνουμε. Τώρα, σε σχέση με τον κανονισμό του 1996, τι είναι το καινούριο. Είναι ότι εμεί θέλουμε μια διαδικασία πιο διάφανη όλα τα δεδομένα τα οποία φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτονται από το απόρριτο. Η Κομισιόν, το Συμβούλιο έχουν πρόσβαση, εμείς δεν τα δημοσιεύουμε αυτά τα στοιχεία. Δεν γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτά με τους εμπλεκόμενους. Προτείνουμε μία δημοσίευση που να αφορά συγκεντρωμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά στοιχεία δηλαδή. Δεν θέλουμε να δημοσιεύουμε στοιχεία για τη μία την άλλη επιχείρηση, ούτε είναι εμπορικό ο σκοπός. Σίγουρα τίθεται θέμα προστασίας δεδομένων. Αυτό θα φροντίσουμε να καλύψουμε, γι' αυτό και δεν δημοσιοποιούμε τις πληροφορίες που παίρνουμε. Αυτό που θέλουμε όμως είναι να μπορούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτικά και με την ε, Κοινωνική Οικονομική Επιτροπή να συζητάμε. Κάθε δύο χρόνια, όπως σας είπα, αυτό προτείνουμε. Γιατί έτσι μπορούμε να δούμε κατά πόσο οι υποδομές, έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί στην Ευρώπη, ανταποκρίνονται στους πολιτικούς στόχου. ναι ή όχι. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκέρεκ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό ότι είναι χρήσιμο να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι μπορούμε καλύτερα να οργανωθούμε και καλύτερα να σχεδιάσουμε την ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική. Οι τελευταίες μας εμπειρίες από τον Ιανουάριο που μας πέρασε δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αποδεικνύουν ότι είναι καλύτερα να είμαστε ενημερωμένοι παρά να οδηγούμεθα σε κρίσεις όπως αυτή με το φυσικό αέριο που είχαμε τότε. Οπότε η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλά κάνουν που ετοιμάζουν αυτό το νέο σχέδιο κανονισμού. Θα αντικαταστήσει το προηγούμενο κείμενο που είχαμε στη διάθεσή μας και το οποίο δεν είναι πια καλό. Γιατί μιλάμε για βιοκαύσιμα, μιλάμε για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Αρχίζουμε, δηλαδή, να βάζουμε και ορισμούς, πράγμα το οποίο παλιά δεν γινόταν καθόλου. Αλλάζει και... Αλλάζουν και οι τιμές, οι ελάχιστες τιμές. Μιλάμε και για τις δυνατότητες αποθήκευσης φυσικού αερίου, για ελάχιστα όρια κιλοβάτ διαφορετικά από αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Όμως πάνω απ' όλα είναι αναγκαίο να ασχοληθούμε με τις ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό το κείμενο όμως πιστεύω ότι πρέπει να συμπληρωθεί σε δύο σημεία. Στο σημείο 2 πρώτα απ' όλα που υπάρχουν οι ορισμοί. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν αναγκαίο να συμπληρώσουμε τις παραμέτρους τεχνικής φύσεως που χρησιμοποιούνται. Για μένα αυτό θα ήταν αναγκαίο γιατί έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Στη συνέχεια υπάρχει ένας ορισμός των διασυνδέσεων Εδώ λείπει όμως ένας ορισμός που θα ήταν πολύ χρήσιμος, ιδιαίτερα στην πρόσφατη κρίση που είχαμε με το φυσικό αέριο. Έπειτα, για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Όταν μιλάμε για προϊόντα Όταν μιλάμε λοιπόν για τη δίληση και εδώ χρειάζεται ένας ορισμός. Στο άρθρο 6 επίσης μιλάμε για την δημοσίευση ε, συγκεντρωτικών στοιχείων. Ίσως εδώ φοβόμαθα ότι με τη συγκέντρωση, μάλλον αποφύγουμε τη συγκέντρωση, δεν ε, προστατεύουμε το εμπορικό απόρριτο. Σε κάποιες χώρες μπορεί να πρόκειται για ένα και μόνο εργοστάσιο. Παλιά αναφέραμε ουσιαστικά μια συγκεκριμένη εγκατάσταση και αυτό βέβαια πλήττει τον ανταγωνισμό. Η κυρία Χόλ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Και συμφωνώ μαζί τους για το ότι Όντως πρέπει να έχουμε μια ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική και αυτή μπορούμε να την έχουμε μόνο αν έχουμε πληροφορίες για τις ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη. Σωστά. Οπότε το Κοινοβούλιο θα στηρίξει τον κανονισμό αυτό. Ιδιαίτερα θα λάβουμε υπόψη και τις αλλαγές με την που από ό,τι φαίνεται επικύρωση θα έχουμε τις συνθήκες της Λισαβόνας. Όμως είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι στην πράξη θα λειτουργεί αυτός ο νέος κανονισμός και ότι θα είναι όσο γίνεται πιο χρήσιμος. Έρχομαι λοιπόν σε κάποια σημεία στο σχέδιο κειμένου και στα σχόλια που έκανε μόλις τώρα η Επιτροπή. Στην αρχική αξιολόγηση αντικτύπου λέει ότι τα κράτη-μέλη δεν συμμορφώθηκαν σωστά με τον παλιό κανονισμό του 1996 και δεν έδιναν τις πληροφορίες που έπρεπε. Αναρωτιέμαι λοιπόν, η Επιτροπή μπορεί να μας εξηγήσει ε, γιατί πιστεύει ότι ο νέος κανονισμός ε, θα έχει καλύτερη ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη. Τα εμπορικά ευαίσθητα θέματα τα ανέφερε και ο κύριος Γκέρεκ και η Κομισιόν. Έπειτα, κατά πόσο τα συγκεντρωτικά στοιχεία μπορούν παρόλα αυτά να αποκαλύψουν ε, μυστικά για επιχειρήσεις των κρατών μελών. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είχαν εκφραστεί ανησυχίε στην Επιτροπή από τις διάφορες πλευρές. Γι' αυτό και το Συμβούλιο δουλεύει πάνω σε αυτό κανονισμό. Οπότε θέλω να ξέρω τα κράτη-μέλη τι γνώμη έχουν γι' αυτόν. Τώρα το θέμα τώρα της διπλής ε, παρουσίασης δεδομένων των επικαλύψεων μερικές φορές απαιτούνται από την νομοθεσία. Σίγουρα θέλουμε να αποφύγουμε περί το γραφειοκρατικό άχθος, όμως μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση. Γι' αυτό θα ήθελα η Επιτροπή να παρουσιάζει έναν πίνακα όπου εξηγούνται εκεί οι απαιτήσει. Δηλαδή, τι ζητάνε από τα κράτη-μέλη, τι πληροφορίε θέλουν. Και έτσι ο κόσμο να μπορεί να καταλάβει με μια μέσα σε ένα πίνακα τι πληροφορίε πρέπει να δίνει. Και πάλι τώρα, όσον αφορά την ισχύ της Λισαβόνας, υπάρχει λοιπόν άρθρο που αναφέρεται στην πολιτική μας αυτή. Ποιο θα είναι τελικά το άρθρο στο, το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή ως νομική βάση. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση κυρίας Χαουλ όσον αφορά τις επιπλέον υποχρεώσεις. Καλό θα ήταν να έχουμε ένα έγγραφο, μια, ένα κατάλογο αυτών των επιπλέον υποχρεώσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σπίτε Χόφερ. Εγώ θα δώσω το λόγο στο σκιώδη εισηγητή, τον κύριο Ζαντό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσία της. Στηρίζουμε και εμείς την ιδέα αυτή μια κοινή ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη. Έχω κάποιες ερωτήσεις και κάποιες παρατηρήσεις. Στο έγγραφο βλέπουμε να μιλάτε για διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις, τους ρυθμιστές κλπ. Θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα Γι' αυτό οι διαβουλεύσεις περιλαμβάνουν και την τοπική αυτοδίκηση που παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στον τομέα των ενεργειακών υποδομών. Επίσης υπάρχουν διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα, με άλλους παράγοντες της ε, κοινωνίας των πολιτών. Αλλά κυρίως το θέμα της διαφάνειας με απασχολεί. Και τα ακούσαμε ήδη ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το τελικά ε, αυτό το απόρριτο που εσείς μας λέτε για τα εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία. θα μπορέσει να γίνει ανοιχτή συζήτηση για τις επιλογές τις ενεργειακές τις οποίες θα καταλήξει η Ευρώπη. Από το έγγραφο αυτό βγαίνει ένα πολιτικό μήνυμα όσο να είναι, για το τύπο ενέργειας που θέλουμε να έχουμε. Μιλάμε πολύ για ε, τα στερά. Μιλάμε πολύ για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, υδρογονάνθρακες κλπ. Αλλά δεν επιμένουμε αρκετά σε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει, δηλαδή μια νέα ενεργειακή πολιτική που να συμπεριλαμβάνει ευφύ δίκτυα διανομής με μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας. από τις πληροφορίες που λέτε εσείς ότι θα συλλέγουμε δεν έχουμε τίποτα ούτε για τα δίκτυα διανομής ούτε για τις μικρές μονάδες παραγωγής. Πριν συζητούσαμε για την οικολογική καινοτομία και είδαμε ότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την οικολογική καινοτομία είναι στα κτίρια. Τον έχουμε δηλαδή κτίρια που να καταλώνουν μηδέν ενέργεια ή τέλο πάντων να είναι περιβαλλοντικά θετικά. Οπότε δεν θα έπρεπε να έχουμε και τέτοιου είδου πληροφορίες για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση για τις ενεργειακές υποδομές. Είπε η Επιτροπή ότι πρέπει να ξέρουμε και τι εμπόδια υπάρχουν για επενδύσεις, ας πούμε η πρόσβαση στις πιστώσεις. Οπότε σε αυτό το κείμενο, γιατί να μην βάλουμε και στοιχεία για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό, πέρα δηλαδή από τα τεχνικά στοιχεία που θα ζητάμε για τις ενεργειακές υποδομές, να ζητάμε και πληροφορίες για την χρηματοδότηση αυτών των υποδομών. Τέλος, πιστεύουμε ότι λείπει κάτι σημαντικό. Είναι αποτελεσματικότητα, η ενεργειακή απόδοση δηλαδή των υποδομών αυτών. Γιατί αν ο στόχος μας είναι να έχουμε την πιο αποτελεσματική ενεργειακά οικονομία, με εκπλήσει που δεν βλέπω κάτι για ένα σύστημα το οποίο να μας επιτρέπει να αξιολογούμε επιμονή μου βάσεω στην ενεργειακή απόδοση των ίδιων των ενεργειακών υποδομών. Ευχαριστώ. κολύγε Μαρινέσκο. κύριος Μαρινέσκο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και να ρωτήσω και μερικά πράγματα. Στην, ε, στο σκεπτικό αναφέρεται το θέμα της ενεργειακής αγοράς. Στο σχέδιο κανονισμού όμως δεν αναφέρεται το παρατηρητήριο καθόλου. Οπότε, για πείτε μας, οι πληροφορίες τελικά από πού έρχονται. θα έπρεπε να πηγαίνουν στο παρατηρητήριο πληροφορίες. Και μάλιστα στο σκεπτικό λέει επίσης ότι το παρατηρητήριο και η Κομισιόν θα κάνουν την ε, ανάλυση τελικά για να ξέρουμε τι προοπτικές υπάρχουν στον ενεργειακό τομέα. Πουθενά όμως δεν λέει πού θα πηγαίνουν οι πληροφορίες αυτές Ποιο θα τις παίρνει μελλοντική υπηρεσία, ενεργειακή, αυτοί θα κάνουν την ανάλυση. Έπειτα, τι εννοείται με το πολιετές πρόγραμμα επενδύσεων στις ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρόθεση. Η στόχοι. Έπειτα. Εσείς ζητάτε στοιχεία. Ένα ενεργειακό πρόγραμμα μπορεί να κρατάει 10 χρόνια. Πότε θέλετε να σας στέλνουμε αυτά τα στοιχεία. Στην αρχή, όταν γίνεται η μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος, όταν είναι έτοιμο το τεχνικό σκέλος, όταν ξεκινάνε οι επενδύσεις, πότε ακριβώς. Ένα απλό παράδειγμα, το Ναμπούκο. Θα ενημερωθείτε για αυτό το πρόγραμμα του 2006 ή όχι. Έπειτα μπορεί να υπάρχουν και επιχειρήσεις που επενδύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδύσεις αυτές όμως μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτές τις επενδύσεις θα πρέπει να δώσουμε στοιχεία ή όχι. Έπειτα στον κανονισμό, το είπε εξάλλου και η Κομισιόν αυτό, ότι η Επιτροπή θα δημοσιοποιεί συγκεντρωτικά στοιχεία. Πρόκειται όμως για πολύ ε, λεπτά δεδομένα, ευαίσθητα, απόρριτα πολλές φορές και αυτό κινδυνεύει να δημιουργήσει προβλήματα. Πώς θα διασφαλίσετε λοιπόν το απόρριτο των ε, δεδομένων αυτών. Ευχαριστώ. κύριος Μπιτικόφ. Δύο ερωτήσεις έχω προς την Επιτροπή. Πρώτον, δεν μπορούμε απλώς να συγκρίνουμε στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες. Εδώ πρόκειται περί μιας πολιτικής δυναμικής, την οποία θέλουμε να απελευθερώσουμε. Τι είδους πολιτική δυναμική επιθυμεί να δημιουργήσει η Επιτροπή με αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κοινή συλλογική ευθύνη για αυτήν την υποδομή. Και ούτε μπορεί κανείς να συσσωρεύσει διάφορα εθνικά προγράμματα και συστήματα και να μιλήσει μετά για ευρωπαϊκές πρόπτικες. Γιατί αλλιώ δεν υπάρχει δυνατότητα δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικό στον τομέα της ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε να υπάρξει παραδείγματος χάρη ένας φορέας, ένας οργανισμός όπως για την πυρηνική ενέργεια του Euratom είτε μια πραγματική συνεργασία που να οδηγήσει σε κοινή πολιτική δράση. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι συγκεντρώνονται πληροφορίες χωρίς να υπάρχει δυνατότητα δράσης κοινή. Ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για την επιλογή των εργαλείων και για την ε, συμφωνία με άλλες ρυθμίσεις. Το έγγραφο αναφέρει 8 διαφορετικά κείμενα, όπου είναι οι διατάξεις που είναι στην ανακοίνωση για την ενεργειακή υποδομή, κανονισμού και οδηγίε, Μήπως θα μπορούσαμε να προστεύσουμε κάποια τα πράγματα έτσι ώστε οι χρήστες του κοινωνικού δικαίου να έχουν ένα κείμενο για το ίδιο θέμα και ο κανονισμό είναι το σωστότερο εργαλείο. στις εξηγήσει αναφέρεται κανονισμό διότι αναθεωρείται ο κανονισμός. Θα πρέπει όμως να πούμε στα εργαλεία γιατί χρησιμοποιείται ο κανονισμός. Και όχι με μόνο το επιχείρημα ότι μπορούμε να αναθεωρήσουμε έναν παλιό κανονισμό. Για τη δημοσίευση των πληροφοριών τώρα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ορισμένε πληροφορίε στρατηγικού εμπιστευτικού χαρακτήρα τελικά δεν θα δημοσιευτούν γιατί μπορεί να υπάρχει κίνδυνο για ορισμένου στην περίπτωση αυτή. Τέλο, φαίνεται ότι δεν προβλέπεται καμία κύρωση. Τι συμβαίνει, τι θα συμβεί μάλλον αν οι φορεί δεν ε, σεβαστούν και δεν τηρήσουν τι υποχρεώσει του. Μπάλσον. Θα ήθελα η Κομισιόν να μας απαντήσει στο εξής ερώτημα. Ποια είναι η σωστή ερμηνεία. Άκουσα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά δεν κατάλαβα καλά. Αν συγκρίνουμε αυτά που λένε τα έγγραφα που έχουμε πάρει με αυτά που ακούσαμε, Μιλάμε για ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής που είναι η αποδοτική χρήση της ενέργειας αλλά και η παραγωγή της ενέργειας σε πιο περιορισμένο πλαίσιο. Διάβασα τα κείμενα και κοίταξε ιδιαίτερα τους ορισμούς. Για ποιες μονάδες μιλάτε, μεγαβάτ, όταν μιλάτε για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τι είδος δυναμικό έχετε κατά νου. Τι θέλετε να ρυθμίσετε σε όγκο με, τις, με, με το μέτρο αυτό. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά. Θέλουμε οι φορείς να παίρνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και να υπάρχει και προβλεψιμότητα για τον καρδιασμό των φορέων για να μπορούν να προσαρμόσουν τις επενδύσεις τους, την βιομηχανική τους πολιτική στις μελλοντικές ανάγκες. Εγώ με βάση τα έγγραφα αυτό δεν το πολύ κατάλαβα. Γιατί συζητάμε. Ήθελα να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι που από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν στο κείμενο. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις έγιναν. Και εγώ έχω μια ερώτηση. Δεν κατάλαβα καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις ήδη στους κανονισμούς, στις οδηγίες. Γιατί δεν τα συγκεντρώνουμε όλα αυτά, αλλά δημιουργούμε άλλη μια διαδικασία υποχρεώσεις. Και ακούσαμε από τον ε, Επίτροπο Φερχόγγεν ότι όλη η άχρηστη ρύθμιση και νομοθεσία θα πρέπει να πάψει να υπάρχει. Μπορώ να σας κάνω την ερώτηση και αλλιώς. Τι από όλες αυτές τις ρυθμίσεις και υποχρεώσεις που υπάρχουν θα καταργηθούν. Και θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Πολλές ε, ερωτήσεις απαιτούν πολλές απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά, γιατί έχω προετοιμάσει το κείμενο στα αγγλικά. Ξεκινάμε με τις θεσμικές ερωτήσεις. Και αν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο παρατηρητήριο της αγοράς και το παρατηρητήριο της Κομισιόν για την ενέργεια. Όχι. Το παρατηρητήριο της αγοράς για την ενέργεια είναι στη Γενική Διεύθυνση ΤΡΕΝ, δηλαδή είναι κομμάτι της Κομισιόν. Δεν είναι χωριστή υπηρεσία. Πάντως το Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστηρίζει τη θέση ότι ένα παρατηρητήριο παρακολουθεί το τι γίνεται γενικά σε όλο το ενεργειακό τοπίο της Ένωσης. αυτό κάνουμε και εμείς. Δεν εξειδικευόμαστε στον άνθρακα ή στην αποδοτική χρήση της ενέργειας ή της ανανεώσιμας κοιτάμε πώς λειτουργεί η δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς και ποιες είναι οι μελλοντικέ εξελίξεις για την υποδομή, παραδείγματος χάρη. Ρωτήσετε γιατί επιλέξαμε κανονισμό. Στηρίχαμε στο άρθρο 281 και 187 της Ευρατόμ διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλη νομική βάση ή άρθρο της συνθήκης. Γι' αυτό ο κανονισμός του 96 και αυτός στηρίζεται σε αυτά τα δύο άρθρα. 284 που η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται από τα κράτη-μέλη για να κάνει τη δουλειά της και το 187 για να καλυφθεί και ο ηλεκτρισμός που παράγεται από την πυρηνική ενέργεια. Άλλο αυτό και άλλο η πρόταση κοινοποίηση όπως προβλέπει η συνθήκη Ευρατόμ. Όταν ένας φορέας σκοπεύει να κάνει ένα νέο πυρηνικό σταθμό, πρέπει να το αναφέρει αυτό στην Κομισιόν που γνωμοδοτεί. Αυτό γίνεται μία και έξω. Η Κομισιόν δεν μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται όσον αφορά καθυστερήσεις και λοιπά στην φάση κατασκευή. Σωστά υπόθηκε και γι' αυτό σας να κοιτάξετε την έκθεση αξιολόγησης. Η κυρία Χόλ το ανάφερε, παράρτημα 3. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές υποχρεώσεις για αναφορά σε διάφορα σημεία του κοινωνικού δικαίου. Το πρόβλημά μας είναι είτε το έγκαιρο της υποβολής αυτών των πληροφοριών, σας ανάφερα τη συνθήκη Ευρατόμ, που γίνεται μία φορά στη ζωή ή ή μπορεί να γίνεται με εντελώ άλλους ορισμού. ή μπορεί να γίνεται σε ένα χρονικό πλαίσιο που εμείς θεωρούμε σκόπιμο. Υπάρχουν όμως νομοθετήματα, ιδιαίτερα πρόσφατα, που συνηγορούν υπέρ της ιστορικής εξέλιξης της πολιτικής για την ενέργεια με τις επιταχύνσεις που γνώρισε στην Ευρώπη. Αυτό δεν το αγνοούμε, το λαμβάνουμε υπόψη. Αυτό που προτείνεται και εφαρμόζεται στο τρίτο πακέτο εσωτερική αγορά, τα προγράμματα επένδυσης για τα δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου. Γι' αυτό προτείνουμε τον κανονισμό για να αποφύγουμε διοικητικά βάρη αντί να ζητάμε με οδηγία μία φορά, περιμένουμε, σε επαφή φυσικά με τους τα ευρωπαϊκά συστήματα, οι φορείς που λειτουργούν στα συστήματα αυτά, θα περιμένουμε να δούμε τι θα μπει σε ισχύ ή μετά από ένα χρόνο θα πάρουμε τις πληροφορίες αυτές και μετά θα ζητήσουμε, θα ρωτήσουμε μάλλον τις κυβερνήσεις. Συμφωνείτε με αυτά που μας λένε οι μεταφορείς της ενέργειας. Αν η... και ανάλογα με την απάντηση θα θεωρήσουμε ότι έληξε η διαδικασία. Ωστόσο σας επισημαίνω ότι επειδή αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέλιξη τα προγράμματα αυτά και συζητάμε ακόμα το χρειάζονται αυτό τον κανονισμό σε δίκτυα ασφαλεία, γιατί ω TSO θα πρέπει να ξέρει κανείς για να προσαρμοστεί το δίκτυο στι μελλοντικέ ανάγκες πρέπει να ξέρει τι δυναμικό προβλέπεται, τι προγραμματίζεται. Και αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι φορείς δίνουν μάχες για να καταλάβουν ε, τι προγραμματίζεται για το μέλλον όσον αφορά την παραγωγή, ε, το δυναμικό παραγωγής ή μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Αναντίθετα, κυβερνήσεις που έχουν τις διοικητικές πληροφορίες όσον αφορά τις άδειες που εκδίδονται για κατασκευή σταθμών κλπ. Και μην ξεχνάμε και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και επίπεδα. Αν, η χώρα, γίνει λοιπόν σε αυτό το επίπεδο επικύρωση, με αξιολόγηση και επικύρωση των καλύτερων συστημάτων μεταφοράς, διότι αυτό που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να κάνουν την πιο καλή εκτίμηση, τίποτε παραπάνω. Μια εκτίμηση μόνο. Γιατί το πακέτο της εσωτερικής αγοράς δεν είναι τόσο λεπτομερές και τόσο σαφές για τα θέματα που συζητάμε. Α, λοιπόν, βλέπουμε μάλλον αυτό στο σημείο ως δίχτυα ασφαλείας και θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και μετριοπαθείς. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα Ίσως οι πληροφορίες που θα πάρουμε να είναι τέλειες, όλες οι χώρες να συμφωνήσουν. Οπότε να πούμε αυτό το νομοθέτημα ισχύει μόνο για την ε, υποδομή, για το πετρέλαιο, για τα δηληστήρια, τα βιοκαύσιμα, όχι όμως για τον ηλεκτρισμό και το αέριο. Προς το παρόν δεν ξέρουμε. Σας καλώ λοιπόν να μελετήσετε το παράτημα αυτό της αξιολόγησης επιπτώσεων και να δείτε πώς γίνονται τα δίκτυα των φορέων, πώς επεξεργάζονται τα δεκαετή τους προγράμματα. Περνάω τώρα στην, στον περιοδικό, στο ερώτημα για τον περιοδικό χαρακτήρα. Επειδή αυτού του είδους οι υποδομές ε, χρειάζονται πολλά χρόνια να γίνουν, προτείνουμε να το κάνουμε κάθε δύο χρόνια και όχι κάθε χρόνο όπως έλεγε ο παλιός κανονισμός. Και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και περισσότερη διαφάνεια. Και βλέπουμε ταυτόχρονα πώς εξηγίζονται μελλοντικέ ανάγκες και έτσι εξασφαλίζεται η δυναμική αυτή διάσταση. Να μπορούμε δηλαδή να προβλέπουμε προβλήματα που θα, εμφανιστούν στο μέλλον όσον αφορά την ενεργειακή υποδομή. Υπάρχουν χώρες που αυτό το κάνουν ήδη εθνικά. Αλλά πολλοί άλλοι φορείς, ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ζητείται η γνώμη τους γι' αυτό. Εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να πέσουμε σε αυτό το τόσο χαμηλό επίπεδο όσον αφορά την, την, τις πληροφορίες. Αλλά με διαφάνεια και δημοσιότητα οι πληροφορίες που φεύγουν από τις Βρυξέλλες εξυπηρετούν το εθνικό επίπεδο, διότι καλύπτεται έτσι η ευρωπαϊκή διάσταση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να υπάρχουν ανησυχίε αν ορισμένες περιφέρειες, παραδείγματος είναι καθαρή εισαγωγής ηλεκτρισμού γιατί όλοι στηρίζονται στο ότι ο γείτονα θα βοηθήσει, ότι θα έχει επιπλέον πλεονάζον δυναμικό αν χρειαστεί. Ο εμπιστευτικό χαρακτήρας των στοιχείων και οι στοιχείε που είναι εμπορικά ευαίσθητε. Δεν θέλουμε να δημοσιεύουμε θέλουμε να δημοσιεύουμε συνολικές αθροίσματα πληροφοριών και να μειωθεί το διοικητικό βάρος και για να αποφύγουμε εμπορικά ευαίσθητη πληροφορία να δοθεί στη δημοσιότητα. Ειδικά για κράτη με τα μικρά που ακόμα σε ένα άθροισμα μπορούν να ξεκαθαρίσει κανείς από πίσω ποιος είναι ο συγκεκριμένος φορέας και τα αντίστοιχα νούμερα θα κάνουμε αυτό που κάνουν και τα άλλα θεσμικά όργανα. Δηλαδή, περιφερειακά θα μαυρίσουμε την πληροφορία αυτή και θα δώσουμε ε, σωρευτικές πληροφορίες μόνο για σύνολο νησιών ή για μια μεγάλη περιφέρεια, έτσι ώστε να αποφύγουμε να εκτεθεί με την αρνητική τώρα ένα συγκεκριμένο φορέα. Αποδοτική χρήση της ενέργειας. τη χρήση υποδομών. Αν και είναι λεπτομέρειε βέβαια Το να έχουμε έξυπνα κτίρια όσον αφορά την ενέργεια στην Ευρώπη είναι στοιχείο ζήτησης. Αυτό λοιπόν το καλύπτουμε με το ενεργειακό σενάριο όσον αφορά τις εξελίξεις. Για την υποδομή Πρέπει να πετύχουμε μια καλή ισορροπία. Από τη μια μεριά, σε ποιο επίπεδο η μικροπαραγωγή απαιτεί παροχή πληροφοριών. Από την σκοπιά της Ένωσης προτιμούμε να ε, χρησιμοποιηθεί η επικουρικότητα και η κάθε χώρα με πρόταση δική μας να αποφασίσει ας πούμε μικροπαραγωγή ηλεκτρισμού, άλλοι μπορεί να πάρουν επίπεδο επιχειρήσεων ή πάρουν επίπεδο νοικοκυριών, αν μπορούν να πάρουν αυτές τις πληροφορίες. Μπορούν να γίνουν έρευνες αντιπροσωπευτικές και να δοθούν αυτές οι πληροφορίες στις Βρυξέλλες χωρίς απέτηση κοινοποίησης για μία συγκεκριμένη επιχείρηση. Και έτσι μπορούμε να κρίνουμε και πώς εξελίσσονται οι ενεργειακές υποδομές και με έναν αποκεντρωμένο τρόπο. Συμφωνώ όσον αφορά την αποδοτική χρήση ή την αποδοτική παραγωγή Δεν αρκεί η πληροφορία για, την, για το ονομαστικό δυναμικό, πληροφορίες για την χρήση αυτού του δυναμικού πόσο χρόνο λειτουργεί, τι είδους ενέργεια παράγει ή τι είδους τεχνολογία επελέγει για την αποδοτική χρήση της ενέργειας. Εμείς θα κρίνουμε αν πρέπει να δημοσιευτεί αυτού του είδους η πληροφορία. Πάντως, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμοι στις αρχές σχεδιασμού. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ζητούνται από τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι αρχές κάθε χώρας θα πρέπει να φροντίσουν συγκεντρωτικά να παίρνουν αυτές τις πληροφορίες και να τις μοιράζονται με τις άλλες χώρες. Θα σταματήσω εδώ, γιατί στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι κάπως πρόωρο νομίζω. Πάντως αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε με email. Ή διμερός. Πρόεδρος, ωραία. Ας κλείσουμε το θέμα αυτό. Σας ότι το σχέδιο θα συζητηθεί 2 με 3 Δεκεμβρίου, τροπολογίας 9 Δεκεμβρίου και μπορούμε να, ψηφί... να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε στις 14 Ιανουαρίου αλλά το Δεκέμβριο θα έχουμε ακουράσεις των επιτρόπων λοιπά. Είναι δύσκολος μήνας. Το σημαντικό είναι 2 με 3 Δεκεμβρίου, όπου θα έχουμε την έκθεση και θα υπάρχει δυνατότητα οι ομάδες να καταθέσουν τροπολογίες. Αποφασίζεται έτσι αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Άλλο διάφορα. Όχι. Πέρα τη συνεδρίασεις. Την επόμενη εβδομάδα ξανά εδώ.